Good morning to you all, colleagues. Καλημέρα συνάδελφοι. Μπορούμε να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Άκουσα ότι υπάρχουν μέλη που θα φτάσουν αργότερα γιατί έχουν προβλήματα. Ας αρχίσουμε όμως με το πρώτο θέμα στη μερίσια διάταξη το οποίο είναι η ανακοίνωση μου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών που ξέρετε ότι συνεδρίασαν χτες ε, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αποφάσισαν για τη συνέχεια που δίδεται στις αναφορές σχετικά με τη μετανάστευση να αποσταλεί επιστολή στην Ελληνική Προεδρία και να ζητηθεί ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας ακριβώς για τέτοια θέματα μετανάστευσης. Επίσης, θα ζητήσουμε τα προβλήματα που συνδέονται με τα μεταναστευτικά να ε, γίνουν προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξή μας. Για το δεύτερο θέμα των συντονιστών, αιτήματα για διαδικασίες κατεπηγόντως, αποφάσισαν οι συντονιστές να ε, δώσουν κατεπήγον ε, στις αναφορές εκείνες που ήδη υπήρχε σύσταση για αυτές. Θα σας αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ε, ο κατάλογος για να αποφασίσουμε ποιες από τις αναφορές αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές, θα εγκριθούν τελικά ως κατεπήγουσες και θα υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Σημείο 3. Αποφάσισαν οι συντονιστές να απορρίψουν το αίτημα αυτό. Το ίδιο ισχύει και για το 4. Στο σημείο 5 και 6 οι συντονιστές θέλουν περισσότερη πληροφόρηση και συμφώνησαν με την Προεδρία για την ε, διαδικασία που εγκρίναμε για να ακολουθήσουμε. Για το σημείο 7, το μελλοντικό προγραμματισμό, αποφάσισαν οι συντονιστές να απορρίψουν το αιτήμα της κυρίας ε, Μπελιέ. Το σημείο 8 οι συντονιστές ενέκριναν ε, την ημερήσια διάταξη για την επόμενη ε, συνεδρίαση, ενώ για τα σημεία 9 και 10 οι συντονιστές ε, σημείωσαν και έλαβαν γνώση της πληροφόρησης που έγινε για το ιστότοπο, τη δικτυακή πύλη δηλαδή, και ε, τις διαδικασίες ε, και τις μεθόδους που ακολουθούνται στις εργασίες της Επιτροπής. Στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών διαβεβάστηκε το θέμα της ειδική έκθεσης για το Frontex. Αυτά. Δεν αποφάσισαν τίποτα άλλο συντονιστές από αυτό που σας είπα και νομίζω ότι σας είπα όλα τα θέματα των συντονιστών. Ο Ντέιβιτ μου λέει να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητε της Επιτροπής μας υπήρχε και οικονομική έκθεση και παρακαλώ όλα τα μέλη να λάβετε γνώση ε, αυτής της ενημέρωσης και των εγγράφων που έχουν διανεμηθεί και σχετικά με την οικονομική αυτή διαχείριση. Ποιος ζητεί το λόγο, θέλει κανείς το λόγο για αυτά που σας είπα. Όχι. Μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών. Και τώρα, όπως είπαμε, θα αρχίσουμε ε, πρώτα από την έκθεση του κυρίου Βαλέσα, το 16 ε, δηλαδή, και του δίνω μέσω στο λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Madam uh, Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε το σχέδιο έκθεσης ε, την τελευταία ε, ετήσια έκθεση για τη θητεία αυτήν. Σε αυτή την έκθεση υπογραμμίζουμε τις δραστηριότητες της Επιτροπής του 2013, αλλά πιστεύω ότι η έκθεση αυτή δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο μια σύνοψη των δραστηριοτήτων μας του τελευταίου έτους. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ανασκόπηση ολόκληρης της κοινοβουλευτικής θητείας. Έτσι προτείνω λοιπόν στο κείμενο αυτό να το χωρίσουμε σε τρία μέρη. Το πρώτο θα είναι η σύνοψη των εργασιών της Επιτροπής μας. Η σύνοψη των επιτευγμάτων μας φυσικά θα επικεντρωθούμε στο περσινό έτος, αλλά όπως πρέπει θα παρουσιάσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τα όσα έχουμε κάνει και επιτύχει σε ολόκληρη τη θητεία. Το δεύτερο μέρος που εγώ ονομάζω νέοι ορίζοντες θα περιλαμβάνει συστάσεις και προτάσεις. Σκοπός θα είναι να γίνει πιο ουσιαστική και ε, πιο επιτυχής η δουλειά της ε, Επιτροπής μας. Προτείνουμε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τις Εθνικές Αρχές. Το τελευταίο κεφάλαιο θα επικεντρώνεται στις μεθόδους εργασίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή μας είναι η φωνή των πολιτών. Εδώ μπορούν να αναφέρουν τις ανησυχίες τους και να γίνουν ακουστοί. Εδώ λοιπόν υιοθετούμε ε, εσωτερικούς, το εσωτερικό κανονισμό και ορίζουμε και τους ε, κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βελτιώσουμε τις εργασίες μας. Χρειαζόμαστε σαφείς προθεσμίες για τον κύκλο ζωή των αναφορών. Χρειάζεται η διαδικασία αυτή να γίνει πιο διαφανής και πιο δημοκρατική. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανόνες των διερευνητικών αποστολών. Σκοπός αυτού θα είναι να γίνουν πιο αποτελεσματικές και να διευκολυνθεί η οργάνωσή τους. Ήδη σε μια συνάντηση των ε, σχεδόν εισηγητών κατέληξαμε σε παραγωγικά αποτελέσματα, αλλά δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εργασίες αυτές. Χρειαζόμαστε τις συμβουλές και του Γιούρα. Μαζί με κάποιες επιπλέον τροπολογίες πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή από την παρουσία μορφή Υπάρχει το ζήτημα της μετάφρασης. Συμφωνήθηκε με τους υπόλοιπους συγγητέ ότι θα εργαζόμαστε μόνο στις αγγλικές εκδοχές των κειμένων. Από κατάλαβα η γραμματεία θα παράσχει υποστήριξη σε όποιο μέλος το χρειαστεί εφόσον δεν γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα. Αυτό απαιτείται λόγω περιορισμένου χρόνου και για να επιταχύνεται η διαδικασία εκπόνησης. Έτσι συμφωνήσαμε λοιπόν ότι η αγγλική γλώσσα θα είναι η μόνη γλώσσα εργασίας αυτή τη στιγμή. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 27 Ιανουαρίου. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να εγκρίνουμε το εγγραφό αυτό 10 ή 11 Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε λοιπόν πολύ χρόνο. Αναμένω να ακούσω τα πρόσθετα σας σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να σας ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρευρίσκεται για αυτό το σημείο. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπέκερ. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν ε, τον ε, εισηγητή. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι εκπλήττω πολύ θετικά όσον αφορά το πόσο ολοκληρωμένη, πόσο ε, εντελεχής είναι η ανάλυση στην έκθεση αυτή και ευχαριστώ πολύ πραγματικά τον εισηγητή. 27 του μηνό είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ουσιαστικές ε, ε, τροπολογίες. Ε, περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή τα πιο ουσιαστικά, αν θέλετε, στοιχεία. Ενδεχομένως μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια σημεία, όπως παραδείγματος χάρη την ε, επιτάχυνση της διαδικασίας εδώ στην Επιτροπή, παραδείγματος χάρη η παραδείγματο χάρη η συνεργασία της δικής μας επιτροπής με άλλε επιτροπές εδώ στο Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι ένα θέμα που ενδεχομένω μπορούμε λίγο να συμπληρώσουμε. Λεπτομέρειες όμως ε, θα ήθελα να προτείνω. Επί της ουσίας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιητική η έκθεση και πραγματικά εμείς θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας μέχρι τις 27. Mr. Ο κύριος Ιρασάμπαλ Μπέιτια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλένσα για το έργο του, για την ε, έκθεσή του και για την προθυμία του και το ανοιχτό πνεύμα διαλόγου και διαπραγμάτευσης, όπως φάνηκε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο που είχαμε τη συνάντησή μας όπως είπε και ο κύριος Βαλέσα, δεν είχαμε διερμηνία και δουλέψαμε στα αγγλικά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό επί της ουσίας, αλλά όταν έχουμε μια τέτοια έκτακτη περίσταση όπως είναι το τέλος της θητείας, δεν θα πρέπει στο μέλλον αυτό να παγιωθεί, να θεσμοθετηθεί και να δουλεύουμε μόνο σε μία ή δύο γλώσσες, έστω και οι σκιώδεις το θέμα με τη Γαλλικία το είχαμε ξαναδεί, δεν υπήρχαν τροπολογίες στα Ισπανικά. Υπήρξε και προηγούμενο. Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας τώρα της έκθεσης. Για μας λείπουν κάποια συμπεράσματα έτσι πολιτικής φύσεως περισσότερο. Πολύ καλά ε, όσα έχει κάνει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μου λείπει μια πολιτική διάσταση που θα είχε ενδιαφέρον σε μια τέτοια έκθεση. Για παράδειγμα, αυτό που λέτε, Έχουν αυξηθεί οι αναφορές το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ υπενιχρά τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή μας για να τις διεκπεραιώνει. Και θα πρέπει σε αυτή την έκθεση βαθύτερα να μπούμε στην ανάγκη ε, υλικοτεχνικής υποδομής που υπάρχει για την Επιτροπή Αναφορών αν θέλουμε να είναι η ε, φωνή ε, των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δικτυακή πύλη, ε, αυτό το πόρταλ θα μας βοηθήσει στο διαδικτύο να δουλεύουμε καλύτερα και ελπίζουμε το συντομότερο να τεθεί σε λειτουργία πριν το τέλος της θητείας αυτής που διανύουμε. Να είναι ε, σε λειτουργία. Επίσης, σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να κάνουμε πιο ευέλικτο το θέμα ε, των αποστολών και των επισκέψεων. Δεν ξέρω, κάπως να το μελετήσουμε γιατί είμαστε λίγο ασυνάρτητοι σε αυτές τις ε, διαδικασίες. Και είναι αρνητικό για την Επιτροπή μας. Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες μας οι επισκέψεις. Θα κάνω και τροπολογίες. Ευχαριστώ καταρχήν τον κύριο Βαλέσα και το επικοδομητικό του πνεύμα και τη διάθεση για συμβιβαστικές ε, τροπολογίες και για συζήτηση. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να αρχίσω σημειώνοντας το γεγονός ότι δεν καθόλου ευχάριστο ε, ευχάριστη δυσκολία που υπάρχει να υπάρχουν τα υλικά στις γλώσσες, τις επίσημες της, ε, του Ευρωκοινοβουλίου. Και το πρόβλημα υπάρχει και για τις εκθέσεις, τις επισκέψεις και νομίζω αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα για τη συγκεκριμένη έκθεση που συζητάμε. Ε, κατά τη γνώμη μου θα ήταν μια σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη των κινητοποιήσεων και των αγώνων των εργαζομένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια σημαντική ε, συμβολή αν θέλετε και στο ρόλο της Επιτροπής Αναφορών αν ο κύριος εισηγητής ήταν σε θέση να δώσει κωδικοποιημένα ε, τα ζητήματα που φαίνεται να είχαν απασχολήσει την Επιτροπή μας το χρονικό διάστημα που πέρασε. Δηλαδή, σε ποια ζητήματα επικεντρώθηκε η προσοχή των ανθρώπων, των κοινοτήτων που κάναν αναφορές στην περίοδο που διανέμουν. Πού συγκεντρώθηκε περισσότερο. Ξέρουμε, υπήρχαν ζητήματα περιβάλλοντος, υπήρχαν ζητήματα εργασιακών σχέσεων. Εν πάση περιπτώσει, κάπως κωδικοποιημένα που, ήταν το, το, κύριο βάρος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για το που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, να οδηγήσει επίσης και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σε πολύ μεγάλα προβλήματα αν θέλετε που αφορούν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν και του Συμβουλίου και των Προεδρίων και των Εθνικών Κυβερνήσεων. Τρίτο ζήτημα. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας είναι η καλύτερη σε θέση να κάνει παρατηρήσεις και προτάσεις τόσο για μια σειρά από διρεκτίβες, κανόνες, αποφάσεις της Κομισιόν ή του Συμβουλίου, όσο και για τον τρόπο υλοποίησής τους ε, σε διάφορες χώρες μέλη. Διότι εγώ δεν είμαι της άποψης ότι τα προβλήματα υπάρχουν μόνο στις εθνικές κυβερνήσεις που δεν εφαρμόζουν συγκεκριμένες διρεκτίβες. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και με διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο κατάλληλες και πόσο λύνουν τα προβλήματα. Βέβαια θα μου πείτε ουδέποτε ήταν θέμα αυτό πιο βαθύ ενασχόλησης επιτροπής. Το, το δέχομαι. Όμως Μπορεί να υπάρχουν ορισμένα συμπεράσματα, ορισμένες ε, ε, υποδείξεις που να είναι σημαντικές για το μέλλον. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας, εγώ δεν σύμφωνο με το σημείο 21 στο οποίο αναφέρεται η έκθεση, διότι θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτού που ονομάστηκε ε, το Ευρωπαϊκό Έτος των, Πολιτών υπάρχουν μια σειρά ρυθμίσεις μια σειρά προγράμματα άκρος επικίνδυνα και άκρος αντιδραστικά. Όπως παραδείγματο χάρη ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται και στην Ελλάδα, στα σχολεία, που επιδιώκει το ξαναγράψιμο της ιστορίας και την εξίσωση του κομμουνισμού με τον ναζισμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, τέτοιου είδους προγράμματα έχουν μεγάλη ε, συμβολή, αν θέλετε, στην αναγέννηση ε, ρατσιστικών, φασιστικών και νοφασιστικών κινημάτων ε, στην Ευρώπη που όλοι μας διαπιστώνουμε σε πολλές χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γκουράκη. Καλώς ορίζω τον συνάδελφο Τζαλέσκι που αντικαταστά την συνάδελφο Κολάσκα Καπομπίνσκα που εγκατέλειψε αυτή την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πολύ υψηλό επίπεδο καθήκοντα. Για να επανέλθουμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Βαλέσα, να ευχαριστήσω τα μέλη που μίλησαν και συνέβαλαν με τις απόψεις τους. Αυτές οι απόψεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τροπολογιών που θα μοιραστούν και θα κοινοποιήσουν στον κύριο Συγητή, τον κύριο Βαλέσα. Ειδικότερα για το ζήτημα που μόλις ε, περιέγραψε ο συνάδελφος ο κύριος ε, το θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο να εμβαθύνουμε την ένδειξη για ε, τομείς αρμοδιότητας ε, για τις αναφορές. Ε, συνήθως κάνουμε κάποιο διαχωρισμό ανά ανατομής αρμοδιότητας, αλλά η δική σας πρόταση από ό,τι κατάλαβα και ελπίζω να γίνει τροπολογία, υποδεικνύει μια οδό μεγαλύτερης επισήμανσης ε, ε, ομάδων πολιτών που στρέφονται προς, την, ε, προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την φύλαξη προγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ε, θα αναπτυχθούν διαφορετικά μοντέλα στις διάφορες χώρες, διότι στη δική μου χώρα, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν, από όσο γνωρίζω, προγράμματα ενημέρωσης ε, με όραμα τέτοιου τύπου. Και αυτό πιστεύω είναι κάτι σημαντικό, ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι για να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τις ε, δράσεις πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας ε, και για να δώσουμε απόψεις για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που μπορεί να οδηγήσουν ε, στην οικοδομήση μιας πραγματικής ε, ευρωπαϊκής κουλτούρας. Δίνω το λόγο στο συνάδελφο κύριο Βαλέσα για να ολοκληρώσει για αυτή την έκθεση. Thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις της. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Όσον αφορά τα σχόλια του κυρίου Αγκουράκη. Ναι, τα περισσότερα πόσα είπατε αναφέρονται στην λογική σκέψη λάμδα, L και στο σημείο 5. Ε, με μεγάλη χαρά βεβαίως θα περιμένω και τις προτάσεις σας, τις τροπολογίες σας και σαφώς και υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί ο κείμενο προς την κατεύθυνση στην οποία προτείνεται. Εγώ πραγματικά θεωρώ πάρα πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι να ανταλλάξουμε απόψεις στα αγγλικά. Αυτό δυσκολεύει την εργασία μας και ελπίζω πραγματικά ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση ε, όσον αφορά την εργασία σε αυτήν την Επιτροπή στο μέλλον. Φυσικά επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι αναφορές. Για τα συμπεράσματα, ναι, βεβαίως περιμένω τροπολογίες από εσάς και το θέμα των τεχνικών αν θέλετε, θεμάτων θα πρέπει και η Επιτροπή να διαθέτει τη δυνατότητα να ανατρέχει σε ε, εμπειρογνώμονες και βεβαίως εδώ θα πρέπει να βασιστούμε όπως το κάνουμε εξαλλού και στη γραμματεία μας. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα βελτιώσουν την εργασία μας και για τις διερευνητικές ε, αποστολές εδώ ενδεχομένως θα πρέπει να ξαναδούμε τους κανόνες ε, που αφορούν την σύσταση αυτών των ε, αποστολών. Σας ευχαριστώ όλους ε, για τις προτάσεις σας, για τη συνεργασία σας και περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία τις τροπολογίες σας. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κύριο Βαλέσσα, να προσθέσω κάτι που παρέλειψε προηγουμένως. Όλες οι παρατηρήσεις ε, που μας επισημάνθηκαν και αυτές που διατυπώθηκαν από τον συνάδελφο κ. Μπέκερ ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσες ε, και πρέπει να τις κοινοποιήσουμε σε όλους. Αλλά θέλω να λάβουμε υπόψη ότι για την παρουσίαση υποβολή τροπολογιών για τις εργασίες αυτής της Κομισιόν φέτος το 2013 πρέπει να δούμε τα νούμερα αν ε, και σημαντική αύξηση των αναφορών που υποβλήθηκαν σχεδόν 10.000 ε, αναφορές υποβλήθηκαν κατά τη θητεία και αυτό σίγουρα έχει κάποια αξία δείχνει ότι έχουμε υψηλές επιδόσεις θεωρώ ότι αυτό αντικειμενικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να συνεχιστεί μια κοινή προσπάθεια βελτίωση των δραστηριοτήτων μα, ώστε να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στου Ευρωπαίου πολίτε. Εδώ κλείνουμε το σημείο με την εκθέση του κ. Βαλέσα. Ο συνάδελφο ε, κ. Σαλαβράκο, ε, που έπρεπε να ασχοληθεί με το επόμενο σημείο, χρειάστηκε να μα εγκαταλείψει για μια ψηφοφορία σε μια άλλη επιτροπή. Περνάμε λοιπόν ε, στο σημείο 17 που αφορά την έκθεση που είχε ανατεθεί στον συνάδελφο τον κύριο Σαλαβράκο μέσα στα επόμενα 30 λεπτά. Περνάμε λοιπόν στην έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα. Τον λόγο έχει ο αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιστρέφουμε σε αυτό το θέμα της έκθεσης για την Ελλάδα Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχαν στην αποστολή αρχής γενομένης από τη Γραμματεία χωρίς καμιά αμφιβολία η αφοσίωση, το έργο ε, και της Ναταλία και του Ντέβιτ Λόου ήταν εκ των όνου Κάνεφ για την εκπόνηση και του εγγράφου αυτού. Ε, μπορεί να είναι εκτενέστατο, από τα πιο εκτενή έγγραφα ε, που παρουσιάστηκαν ποτέ στην Επιτροπή μας, αλλά το απαιτούσε και το ταξίδι και οι αναφορές. Το λέω αυτό διότι ήταν πολύ εντατική η δουλειά μας και το ταξίδι ολόκληρο και οι επισκέψεις ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω εκτός από τη γραμματεία ε, και τους συναδέλφους ε, που είχαν την καλοσύνη να έρθουν στην αποστολή αυτή για να πάμε μαζί σε όλα αυτά τα μέρη της Ελλάδας. Μπαλτίνη, η κυρία Παλιαδέλη, ο κύριος Χουντής και ο κύριος Αλαβράκος και νομίζω ότι μπορούμε τουλάχιστον να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας διότι καταφέραμε επί τόπου στην Ελλάδα να δούμε κάποια πράγματα και επίσης κυρία Πρόεδρε είμαστε ικανοποιημένοι και από την έκθεση που ερχόμαστε εδώ να παραδώσουμε σήμερα. Αρχίζει με μια εισαγωγή έκθεση αυτή για ποιο λόγο πήγε αυτή η αποστολή. Έχουμε αναφορές ε, στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια και σε όλο αυτό το διάστημα προετοιμάζαμε αυτή την αποστολή. Μετά την εισαγωγή έχουμε το κεφάλαιο που αφορά την επίσκεψη αυτή καθ' αυτή και διαιρείται σε τρεις ε, μέρες, σε τρεις αποστολές, στην Αττική, Αθήνα και Γραμματικό. Είδαμε τις εθνικές αρχές ε, στην πρωτεύουσα της χώρας αλλά και τις περιφερειακές και τοπικές και τους ε, αναφέροντες που ήταν οι πρωταγωνιστές μας, ε, πώς αλλιώς θα γινόταν. Τη δεύτερη μέρα πήγαμε στην Αρκαδία και στην Αττική πάλι, ε, Μεγαλόπολη και Φιλή και την τρίτη μέρα που επίσης αναγράφεται στο έγγραφο αυτό, πήγαμε στη Θεσπρωτεία και στην Ίσο Κέρκυρα, όπου είδαμε επιτόπου και πάλι τα προβλήματα που συνδέονται με τις αναφορές που είχαμε λάβει εδώ. Επίσης βήγαμε στο Καρβουνάρι και τη Λευκήμη, δηλαδή συγκεκριμένα τα και Κέρκυρα. Όπως όλα τα έγγραφα αγαπητοί Πρόεδρε, νομίζω ότι το ζουμί είναι στα συμπεράσματα. Εκεί είναι η κεντρική ιδέα και η σπονδυλική στήλη του τι εστί αυτή η ε, αποστολή και τι θα πρέπει να γίνει, τι μελγενέστε ε, στο μέλλον. Αυτό είναι στα συμπεράσματα. Διαβιβάσαμε τα συμπεράσματά μας, 11 τον αριθμό, που ε, οι συστάσεις μάλλον είναι 11, βασίζονται σε διάφορα σημεία ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο για την διάθεση των αποβλήτων στην Ελλάδα, σημασία το πού εγκαθίστανται ηχητά. Ε, επίσης, λέμε ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πάρα πολύ σημαντική και ουσιώδης. Επίσης τονίζουμε το γεγονός ότι η δημόσια ενημέρωση θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να λαμβάνουν γνώση οι πολίτες έτσι ώστε να μπορούν να την αξιολογούν και να κάνουν και τροποποιήσεις στη δημόσια διαβούλευση, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαπιστώσει, μάλλον να το, να το πω θα πρέπει να αξιολογήσει και να θεωρήσει την πολιτική των κοινοτικών κονδυλίων. Τι εννοώ. Θα πρέπει να προσέχει πού πηγαίνουν τα λεφτά, πώς δαπανώνται, αν πιάνουν τόπο, τι τα κάνουν κτλ. λοιπά Και Και επίση θα πρέπει να υπάρχουν κοινωνικά επιστημονικά κριτήρια και κυρίως αυτό που μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει και έλεγχος για τη διαφάνεια στη διαχείριση για όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων Σας είπα τα συμπεράσματα και η συστάση είναι το πιο σημαντικό και σας τα συνόψισα και μετά από αυτά τα σχόλια νομίζω ότι έχει ανοίξει και προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για αυτό το ζήτημα και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε στην επόμενη συνεδρίαση να το ψηφίσουμε με τις ε, τροπολογίες που θα εγκριθούν ως τότε και τα σχόλια που μπορεί να κάνει κάθε συνάδελφος. Με χαρά να τα ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Τρογκάης. Εκ μέρους της Κομισιόν βρίσκεται ο κύριος Κονινιώτης, στον οποίο θα δώσω το λόγο για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή θα ήθελε εδώ να σημειώσει όλες αυτές τις συστάσεις, να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή καθώς και τον εισηγητή. Δεν ξέρω αν θέλετε να εντοπίσουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Ναι, υπάρχουν κάποια στοιχεία που χρειάζονται συζήτηση ενδεχομένω. Euh, euh, Α πάρουμε τι τρει αναφορέ. Όσον αφορά το γραμματικό, όπως είπαμε και στην τελευταία συνεδρίαση τη ε, Επιτροπής αναφορών, έχει συζητηθεί αυτό το θέμα πολλές φορές στο στο ανώτατο κυριωτικό δικαστήριο της Ελλάδας και φυσικά κάποια από τα στοιχεία που περιέχονται στην αναφορά θα πρέπει ενδεχομένως να ε, αναθεωρηθούν. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν παρατηρείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Όσον αφορά το κανονάρι εδώ έχει ξεκινήσει η υπόθεση αυτή, πρόκειται για παραβίαση, έχει ξεκινήσει η διαδικασία και Πρέπει να σας πω ότι στην τελευταία επιθεώρηση που έγινε επιτόπου, το συμπέρασμα είναι ότι ναι, συνεχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες, παρόλα αυτά η κατάσταση σήμερα έχει βελτιωθεί. Γι' αυτό και βεβαίως περιμένουμε τα νέα στοιχεία που απορρέουν από τις επιθεωρήσεις για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Όσον αφορά την Ερμιονίδα, εδώ Βλέπουμε διάφορα σημεία να περιέχει αυτή η αναφορά και θα θέλαμε εδώ να σας επιβεβαιώσουμε ότι και εδώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση και από τις 20 Νοεμβρίου του 2013 έχουμε ε, στείλει μια επιστολή στην Ελλάδα προειδοποιητική και περιμένουμε την απάντηση των ελληνικών αρχών για να συνεχιστεί η διαδικασία, αν βεβαίως αυτό είναι απαραίτητο. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι μετά από την ενημέρωση που έγινε μέσω της Επιτροπής σας στην Εκτελεστική Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αρμόδιο πιλωτικό πρόγραμμα μας έχει ε, δείξει ότι η οδηγία 9383 9883 δεν παραβιάζεται όσον αφορά την ε, ανθρώπινη κατανάλωση. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ναι, υπάρχουν κάποιες υπερβολικές περιεκτικότητες που αναφέρονται κυρίως σε στοιχεία που βρίσκονται στο παράρτημα 1, ιδιαίτερα για την γεύση, για διάφορα βακτήρια και βεβαίως και για το χλώριο. Και βεβαίως ε, εδώ αναφέρομαι στο σημείο C του παραρτήματος 1. Πρόκειται για τιμές τις οποίες ελέγχουμε Υπάρχουν επίσης και στο άρθρο 8 τα διορθωτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ από τις ελληνικές αρχές. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν γίνονται οι επιθεωρήσεις και όταν απαιτούνται να ληφθούν μέτρα από τα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο γίνεται. Τώρα, ό,τι δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1C αλλά στο β του παρατηρήματος 1 και αφορά τα διάφορα, τα διάφορα νητρικά, τον Απρίλιο του 2013 οι έλεγχοι που έγιναν έδειξαν μία σχετικά υψηλότερη τιμή 2 μιλιγκράμμ αναλύτρο, ενώ η οδηγία έχει χαμηλότερες τιμές. Πρόκειται για κάποιες παραβιάσεις οι οποίες βεβαίως εάν παρατηρηθεί ότι επαναλαμβάνονται θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Εάν και εφόσον βεβαίως η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Νομίζω ότι αναφέρθηκα και στις τρεις αναφορές και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση, αυτή την ανασκόπηση. Αναμένω στην επόμενη παρέμβαση κάτι που να επικεντρώνεται περισσότερο στην ε, αποστολή και στα αποτελέσματά της και όχι στο ιστορικό των αναφορών που ούτως άλλως έχουν ήδη ληφθεί στην... και συζητηθεί στην Επιτροπή αυτή ε, παλαιότερα ε, όταν εξετάσαμε τις σχετικές αναφορές. Δίνω το λόγο στο συνάδελφο κ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μετήχαν στην επίσκεψη και βεβαίως τη γραμματεία, τη γραμματεία της Επιτροπής μας γιατί έχει κάνει πολύ συστηματική και υπεύθυνη δουλειά. Πριν μπω στις ε, παρατηρήσεις μου κύριε Πρόεδρε στην έκθεση θέλω αγαπητοί συνάδελφοι να σας αναφέρω ένα πρόσφατο γεγονός που έχει σχέση με αυτά τα θέματα και που όπως σωστά παρατηρήσατε κυρία Πρόεδρο έχει σχέση και το πώς η Κομισιόν, τουλάχιστον με τον αντιπρόσωπό της σήμερα, αντιμετωπίζει τα θέματα. Μετά από επανειλημμένες ερωτήσεις για την περίπτωση του χώρου υγειονομικής ταφής στη Μαυροράχη, άλλη περίπτωση, δεν την επισκεφτήκαμε, παίρνουν την απάντηση, ας την επιβεβαιώσει ο κύριος εκπρόσωπος της Κομισιόν, ότι ξεκινάει η Κομισιόν έρευνα για τη λειτουργία αυτού του χιτά. Ενημερωτικά σας λέω. Θα μας απαντήσει. Είναι επίσημη απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση. Γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Διότι αυτός ο χιτά με κοινοτική χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση, άρχισε να λειτουργεί ως υπερσύγχρονο έργο το 2008 κύριε Έξι χρόνια μετά τη λειτουργία του, τι αποδεικνύεται, ότι έχει πρόβλημα, ο βιολογικός καθαρισμός συγγνώμη, δεν επαρκεί για να διαχειριστούν τα στραγγίσματα, με συνέπεια να επιστρατεύονται διτιοφόρα και να παίρνουν τα στραγγίσματα και να τα πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη στο βιολογικό καθαρισμό με συνέπειες περιβαλλοντικές και οικονομικές κύριε Και οικονομικές Και τι γίνεται τώρα. Εδώ και χρόνια όταν καταγγέλαμε και προειδοποιούσαμε και γι' αυτό το χιτά. Ότι έχει κατασκευαστικά λάθη. Ότι φτιάχτηκε κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που δεν μπορεί. Και εκτός των άλλων, τότε η Κομισιόν ένιπτε, έκανε, πως δεν καταλάβαινε, να το πω έτσι γιατί πήγα να χρησιμοποιήσω μια ευαγγελική ρίση των Ευαγγελίων. Πάω τώρα στην ίδια μας την έκθεση. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε με πιο συγκεκριμένη αποτύπωση αυτών που είδαμε και των στοιχείων και των γεγονότων για τα συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν τεθεί σωστά θέματα και στις συστάσεις περιλαμβάνονται σωστές κατευθύνσεις. Αλλά αυτό είναι ικανοποιητικό διότι διαπιστώνονται ορισμένα πράγματα που πρέπει να επισημανθούν και για τη συνέχεια της υπόθεσης αλλά δεν δίνουν απάντηση και στο συγκεκριμένο στις περιοχές που συναντηθήκαμε, εκεί που πήγαμε τι πρέπει να γίνει. Και εδώ προφανώς υπάρχουν χιτά που βρίσκονται σε λειτουργία και χιτά χώροι υγειονομικής σταθής που βρίσκονται υποκατασκευή. Επομένως η παρατήρησή μου για το συγκεκριμένο θα έλεγα σε αυτούς που βρίσκονται υποκατασκευή και έχουν αποδειχθεί ότι υπάρχουν αστοχίες στις μελέτες και στην κατασκευή, ότι υπάρχει κίνδυνος και ήδη έχουμε διασπάθηση με αυτή την έννοια ευρωπαϊκών κονδυλίων να το αποτρέψουμε. Η περίπτωση του γραμματικού είναι χαρακτηριστική. Έχουν ήδη δαπανηθεί 25 εκατομμύρια, πρόκειται να δαπανηθούν 200, αν είναι ακριβή τα στοιχεία που έχω, προκειμένου να γίνουν τα εργοστάσια και πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα να σταματήσει αυτό το έργο πριν υπάρξουν αυτές οι δαπάνες, από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, και λάθη όσο αφορά την ε, μελέτη, πρόδειλα σφάλματα και προβλήματα τα οποία είδαμε εκεί. Και αναφέρομαι πάλι για το καραματικό, εκεί είδαμε ρέματα. Όσοι επισκεφθήκαμε είδαμε ρέματα μέσα στο χώρο. Το βεβαιώνουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να το γράψουμε στο συμπέρασμά μας. Αν δεν το γράψουμε, τότε δεν μπορεί να στηρίξουμε αυτό το αίτημα ότι εκεί γίνεται λάθος κατασκευή, γίνεται σε λάθος χώρο κατασκευή τέτοιας υγειονομικής, ε, χώρου υγειονομικής ταφής. Ούτως ώστε και η Κομισιόν με σαφήνεια και να τεθεί των ευθυνών να λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Δεύτερο παράδειγμα, το ίδιο και με το καρβουνάρι. Και εκεί πάλι υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουν γίνει απαραίτητες μελέτες. Δεν έχει εξακριβωθεί πού βρίσκεται ο υδροφόρος ορίζοντας και στην περίπτωση του γραμματικού και στην περίπτωση του καρβουναρίου και στην περίπτωση του γραμματικού που είναι υποκατασκευή πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υδρογεωλογικές μελέτες δεν έγιναν και αρνούνται να γίνουν και τις κολυσιεργούν να γίνουν και δεν γίνονται κατάλληλες ούτως ώστε να δοθεί απάντηση σε αυτό το θέμα που σας είπα και το πρόσφατο παράδειγμα με το οποίο ξεκίνησα την τοποθέτησή μου. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι οι αρχές δεν έχουν πάρει υπόψη την οδηγία του 2008 όταν ενέκριναν τις, ή αναθεωρούσαν τις αδειοδοτήσεις. Εν ολίγης, όταν προχωρούσαν δεν έπαιρναν υπόψη την ανανέωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ούτως ώστε να πάρουν υπόψη τους και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία ετίθενται εκεί. Ε, εν πάση περιπτώσει ε, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι κατά βάση το κείμενό μας έχει σωστά συμπεράσματα, δεν έχω καμιά αντίρρηση ως προς εκεί. Οι κατευθύνσεις και οι επισημάνσεις της είναι σωστές. Όμως η, προσπάθειά μας νομίζω ότι πρέπει να γίνει να είναι πιο συγκεκριμένη για τις περιπτώσεις που είδαμε, να είναι πιο συγκεκριμένες και οι προτάσεις μας και οι συστάσεις μας προς την Επιτροπή, προς την ε, Εθνική Αρχή, προς την Επιτροπή, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν, θα έλεγε κανείς, χωρίς παρερμηνίες και θα είναι ένα καλό δείγμα ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η τακτική και όλα αυτά που λέγονται. Η νοοτροπία, η χωροθέτηση, η κατασπατάληση των κοινωτικών χώρων και όλα αυτά που λέγονται υπό τη γενική μορφή να πάρουν συγκεκριμένη μορφή διότι και τελειώνω όπως τα είδαν οι κύριοι συνάδελφοι γύρω από τα προβλήματα αυτά γύρω από τους χώρους αυτούς υπάρχει μια προσδοκία από τον κόσμο που πλήττεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και περιμένει λοιπόν και από την έκθεσή μας μια ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει το πράγμα ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση ή ότι, ότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται τέτοια πράγματα γιατί αυτό που θα ήθελα να σας πω και τελειώνω είναι με αφορμή και το παράδειγμα που σας είπα της Μαυροράχης ενισχύονται τα συμπεράσματα ότι στην Ελλάδα οι μελέτες, οι χωροθετήσεις, οι μελέτες και η κατασπατάληση των κοινοτυπικών πόρων με πολλαπλάσια δυσμενή αποτελέσματα γίνεται με έναν τρόπο όχι αυτόν που συνάδει στις ανάγκες προστασίας του, της, ε, του περιβάλλοντος και της ζωής των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χοντή. Ο κύριος Αγγουράκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, πράγματι αυτή η επίσκεψη ήταν σημαντική στην, Ελλάδα ε, γιατί ξέρετε αυτά τα προβλήματα έχουν γίνει πια εκρηκτικά. Επιπλέον να σας ενημερώσω ότι πέρα από τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει ο κόσμος ε, στην Ελλάδα εμφανίστηκε και το καινούριο της Θολομύχλης λόγω των πολύ ψηλών τιμών του πετρελαίου και του γεγονότος ότι πάρα πολλοί στις μεγάλες πόλεις καίνε πια ακατάλληλα υλικά για να ζεσταθούν τώρα το χειμώνα με φοβερές συνέπειες στην υγεία και στο περιβάλλον. Το λέω αυτό απλά για να σημειώσω <clears throat> ότι γενικά το περιβάλλον στην Ελλάδα χειροτερεύει από την κάθε μέρα που περνάει. Τώρα, για τα δικά μας για την έκθεση. Πραγματικά είναι τεράστια η δουλειά που έγινε από την αντιπροσωπεία και από την ε, γραμματεία της αντιπροσωπείας. Και νομίζω ότι και με, τα, με όσα είδατε και με όσα διαπιστώσατε βγάλετε το συμπέρασμα ότι πράγματι άξιζε τον κόπο αυτή η επίσκεψη. Ε, θα ήθελα όμως ταυτόχρονα να σημειώσω το εξής ότι δυστυχώς παρά τα πολλά στοιχεία και την πολύ κουραστική δουλειά που είδατε, <laughs> είδατε μόνο την κορφή του παγόβου της κατάστασης στην Ελλάδα. Αυτή είναι αλήθεια. Και φυσικά δεν είχε κανείς την απέτηση με μια επίσκεψη και με τις πολύ σημαντικές επισκέψεις που κάνατε να λυθούν όλα τα προβλήματα ή τα προβλήματα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι δυστυχώς τα προβλήματα οξύνονται, πολλαπλασιάζονται και αν θέλετε και με μία έννοια ακόμα και εκεί που πήγατε ή ακόμα και σε αυτά τα, τα σημεία τα οποία ε, τα αναφέρει η έκθεση. Γιατί ξέρετε υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και νομίζω αυτό θα έπρεπε να υπάρχει και ένα συμπέρασμα σε ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε πρέπει να υπάρχει και το θέμα της τιμωρίας ορισμένων οργάνων, ορισμένων επιχειρηματιών, ορισμένων αρχών για πράγματα που δεν εφαρμόσαν. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδου ε, κυρώσει, ούτε καν προτάσει. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα στα συγκεκριμένα. Ε, πράγματι νομίζω ότι στο βαθμό του δυνατού είναι ανάγκη τα συμπεράσματα να είναι πιο συγκεκριμένα για τα σημεία που ε, επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία. Στο βαθμό που μπορεί να συμβεί αυτό. Παραδείγματο χάρη, σα δίνω ένα παράδειγμα που μου κάνει εντύπωση από την έκθεση. Η έκθεση θεωρεί ως ελαφρυντικό στοιχείο για ένα έργο την μαρτυρία ενός μηχανικού που έχει κατασκευάσει κάποιο έργο στο συγκεκριμένο σημείο λέγοντας ότι με τα όσα είπε ο μηχανικός στην, ε, στην Επιτροπή όλα είναι μια χαρά. Ε, αυτό όμως δεν μπορεί να... και, και, και ε, σημειώνεται μαρτυρία, ως, ως τεκμήριο στην έκθεση. Ε, δεν μπορεί ο κατασκευαστής, ας πούμε, να είναι και ο ελεγκτής για το έργο που κάνει. Θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη, εν πάση περιπτώσει, γνωμοδότηση. Δεύτερο, κεντρική σημασία ζήτημα για μας. Ε, επιβεβαιώθηκε και από την τοποθέτηση του εκπροσώπου της ε, Κομισιόν ε, ότι οι καταγγελίες που κάναμε για την κατάσταση της Ερμιώνης είναι σωστές και είναι αληθινές. Βέβαια, ε, πάλι η Κομισιόν ασχολείται μόνο με ένα μέρος του προβλήματος. Για το τεράστιο πρόβλημα των απόβλητων δεν ακούσαμε τίποτα, τα σκουπίδια, του, τους που ξεχυλίζουν στους ε, δρόμους ε, εκεί των, ε, κοινοτήτων και κυρίως θέλω να σας ενημερώσω για το ότι αυτό που είπα και πριν οι διαδικασίες τρέχουν πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Ξέρετε τι έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή. Από την έκθεση είδατε ότι εκεί υπάρχει μια μονάδα, ένα ξενοδοχείο που θέλει να, μια πολυεθνική που θέλει να, να μια μεγάλη μονάδα με γκολφ κτλ. κτλ. Επειδή η μελέτη περιβαλλοντολογικών ε, ε, επιπτώσεων είναι διάτρητη, οι κάτοικοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας να λύσουν το πρόβλημά τους δικαστικά, εν πάση Τι κάνει η Περιφέρεια και η ελληνική κυβέρνηση πριν βγει η απόφαση του, ε, του ανώτατου δικαστηρίου δίνει άδεια κατασκευής της συγκεκριμένης μονάδας. Επαναλαμβάνω, ενώ η, η, η, η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων είναι διάτρητη, έχει προβλήματα, την έχουν καταγγείλει κάτι και έχει πάει στο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχει γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ε, εκρεμεί η απόφαση του Συμβούλιο Επικρατείας για το Μάη φέτος. Πέρσι το Νοέμβρη η κυβέρνηση και η περιφέρεια δίνουν άδεια στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Και έρχομαι σε ένα θέμα γενικότερης νομίζω σημασίας που πρέπει νομίζω να το δούμε σε ορισμένες περιπτώσεις ξέρουμε ότι η Κομισιόν παρεμβαίνει σε ορισμένα έργα με την ολοκλήρωσή τους. Το έχουμε ακούσει και σε άλλες περιπτώσεις. Που είναι πάρα πολύ αργά. Όταν έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση είναι πάρα πολύ αργά και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ε, τέτοια έργα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της φυλής, στην οποία αναφέρεται και η έκθεση, εδώ έχουμε καινούργια προσφυγή των κατοίκων και νομίζω δικαιολογημένα οι οποίοι οι κατοίκοι πολύ σωστά ζητάνε να κλείσει. Να κλείσει αυτή, αυτή η χωματερή. Και δεν είναι μόνο και αίτημα των, των κατοίκων της φυλής, της περιοχής και του συλλόγου. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης της Αττικής βγήκε προχθές και είπε ότι αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα, το 2014 ε, η, η χωματερή της, της φυλής θα ξεχυλήσει. Και λέω, Ποιο αναλαμβάνει την ευθύνη για τους κάτοικου να ζουν σε μια περιοχή η οποία για να αποκατασταθεί όπως λέει πολύ σωστά ε, ε, το πόρισμα της ε, επίσκεψης θέλει 200 χρόνια. Και κλείνω με το εξή. Επειδή κάπου γίνεται λόγος ότι δήθεν για μια συγκεκριμένη περίπτωση κάποιοι δεν θέλανε να, να, να δημιουργηθεί ένα σχητά ε, στην περιοχή τους γιατί θέλουν να, να δημιουργηθεί στην αυλή του γείτονα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Και δεν είναι αλήθεια ούτε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν τεκμηριώνεται ε, πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα και δεν είναι και σωστό γενικά ως αντίληψη, όπως το διαπιστώνει και η, ε, ε, και η έκθεση. Και τέλος, επειδή σημειώνεται ότι οι, οι φορείς, οι εργαζόμενοι προσδοκούν από την Επιτροπή, από τη μελέτη και από τις καταγγελίες της, πρέπει να πούμε ότι οι πολίτες δεν μας χρωστάνε τίποτα. Εμείς τους χρωστάμε. Και μάλιστα ε, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Ευθύνες τεράστιε έχουν στην Ελλάδα διαχρονικά οι κυβερνήσει και του Πάσο και της Νέα Δημοκρατία και συνεχίζουν αυτή την πολιτική, την απαράδεκτη. Ευθύνε υπάρχουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κομισιόν, η οποία γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις και δεν κουνάει το δαχτυλάκι της εάν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμο και αν δεν αντισταθεί και αν δεν αγωνιστεί. Και εμεί τους παροτρύνουμε να είναι ακόμα πιο απαιτητικοί, να αγωνιστούν ακόμα περισσότερο, να παρακολουθούν ακόμα περισσότερα τις, τις εξελίξεις, δεν έχουν δικαίωμα, δεν τους χαρίζει κανείς τίποτα. Πληρώνουν από το ειστέρημά τους, ε, ε ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν τους κοστάει κανένας τίποτα, πρέπει να αγωνιστούν γιατί αυτά τους ανήκουν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ε, Ευχαριστώ το συντάκτη της εκθέσεως και τη γραμματεία για την πολύ καλή δουλειά που κάνανε. Βεβαίως άκουσα και τους συναδέλφους και συμμερίζομαι όλες τις απόψεις τις οποίες εξέφρασαν διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με χώρους στις οποίες διαχειρίζονται απόβλητα και επηρεάζουν δυσμενώς τη ζωή των κατοίκων, την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ε, ιδιαίτερα στη φυλή πρέπει να καταλάβετε ότι είναι μια περιοχή που δεν μπορεί να, υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Με τα επιστημονικά δεδομένα και με τα πραγματικά δεδομένα δεν πρέπει να ζει σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από εκεί άνθρωπος. Μολύνεται. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Ε, από εκεί και ύστερα όμως το θέμα έγκυται στο μέχρι πού νομικά επί τη βάση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μπορούμε να φτάσουμε βλέπω ότι οι συστάσεις τις οποίες και τα συμπεράσματα τα οποία έχει η έκθεση αυτή κινούνται μέσα στα νομικά πλαίσια και φοβούμε ότι οτιδήποτε πάει πέρα από τις συστάσεις αυτές θα παραβιάσει την αρχή της επικουρικότητας διότι η διαχείριση των αποβλήτων ξέρετε είναι θέμα το οποίο εναπόκειται στη διοίκηση των κρατών μελών. Και η άσκηση της διοικήσεως έχει όλα τα, αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα δεν θέλω να το πω ότι είναι η μόνη χώρα που έχει διαφθορά και πίσω από όλη αυτή την ιστορία ε, στείνεται ένα πανηγύρι ε, πάνω στον ανθρώπινο πόνο και όλοι αυτοί οι εργολάβοι και όλοι αυτοί οι, οι υπάλληλοι οι εκείνοι οι οποίοι δίνουν τις δουλειές αυτές έχουν οικονομικά ωφέλη, δυστυχώς. Και φαντάζομαι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ε, πρέπει να το καυτηριάσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα κράτος που ενεργεί, και εγώ έχω μάθει να ενεργώ, πρέπει να πάρει και ορισμένες αποφάσεις τις οποίες δεν μπορεί να το επιτρέψει κανείς. Συνεπώς εγώ θα ήθελα μια καλύτερη ανάπτυξη των συστάσεων στο σημείο 6, 7 και 8 εις τρόπον ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην διαχείριση των αποβλήτων με παρέμβαση της Επιτροπής. Διότι ε, αυτό θα αποτελέσει ίσως ε, και έναν περιορισμό και ένα ανάχωμα στην πάση φύσεως διαφθορά και στην πάση φύσεως ε, κατάχρηση εξουσίας και οικονομικών μέσων που γίνεται σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις. Και θα παρακολουθήσω τον κύριο Ιντρουγάης σε αυτό και μόνο το σημείο, στο 6, 7 και 8, να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση, ε, ξέρει, έχει τον τρόπο, που να φτάσουμε στο όριο που δεν μπαίνουμε μεν στην παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, αλλά λέμε και πέντε κουβέντες παραπάνω να καταλάβουν ότι καταλάβαμε να καταλάβουν και αυτοί κάτω οι πάσης φύσεως τύποι οι οποίοι διαχειρίζονται αυτά τα θέματα ότι καταλάβαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο τα διαχειρίζεται δεν είναι ο πλέον έντιμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you to you. Εγώ σας ευχαριστώ όλους σας. Και τώρα, ορίστε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αφού έχουμε και πολωνική διερμηνία θα μιλήσω πολωνικά. Λοιπόν, ίσως να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο πρώτα. Γενικότερο, πέρα των θεσμικών οργάνων, θα πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ είμαστε εμείς Επιτροπή Αναφορών. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά απλός πολίτης ή κάποιος υψηλόβαθμος, ε, όποιος γνωρίζει την ύπαρξη της Επιτροπής μας μπορεί να απευθύνεται σε εμά. Το είπατε και εσείς Πρόεδρε ότι έχουμε πληθώρα αναφορών που υποβάλλονται, παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερες και χαίρομαι που αυξάνεται ο αριθμός τους. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρόβλημα και μάλιστα δεν μειώνεται αλλά αυξάνεται αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και αλλού. Στο σημείο 8 αναφέρεται αυτό ε, στις συστάσεις για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις χιτά και κτλ. Πώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και με βάση ποια κριτήρια. Και γίνεται λόγος και για τη φωνή των πολιτών. Θα πρέπει να ενημερώνονται οι τοπικές κοινωνίες ε, για την εγκατάσταση στην περιοχή τους ενός χιτά, μια μονάδας ε, ανακύκλωσης αποβλήτων ή λιμάτων σκεφτείτε τι γίνεται με όλα τα πλαστικά ας πούμε ε, που έχετε. Όταν αγοράζεις οτιδήποτε, ένα τηλέφωνο κινητό, ένα ποτήρι, έχεις ένα σωρό πλαστικά σκουπίδια οι ε, ε, κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές πολλές φορές χρησιμοποιούν ε, κοινοτικά κονδύλια για την κατασκευή τέτοιων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαφωνούν με την κατασκευή μιας μονάδας στην περιοχή τους. Θα πρέπει και αυτό να λαμβάνεται υπόψη. Λοιπόν, πώς λύνουμε αυτές τις εντάσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση από τη μια θέλει κάποιος να κατασκευάσει μια μονάδα και από την άλλη έχει τους πολίτες που διαφωνούν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Συνήθως, προφανώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές. Εν πάση περιπτώσει, προσωπικά πιστεύω ότι τα σχόλια του κυρίου Βαλέσα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, μπορούμε να ε, έχουμε κάθε φορά αρκετό χρόνο για διαβούλευση για να συζητούμε και τις συνέπειες. Όπως λέγουν και οι Έλληνες συνάδελφοι, έχουμε καταδείξει τα προβλήματα και έχουμε δει ότι ε, έχει γίνει κακή χρήση κονδυλίων. Έχουν διαχειριστεί κοινοτικέ επιδοτήσεις σε κατευθύνσεις που δεν θα όφυλαν. Δεν ξέρω αν είναι ζητήματα διαφθοράς εδώ ή άλλα κακοδιαχείρισης. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνεται στη φάση του σχεδιασμού μιας μονάδας πριν ληφθεί η τελική απόφαση. Να συμμετέχουν όλες οι πλευρές, να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, ποια είναι τα ωφέλη και ποια είναι ε, τα συμπεράσματα και οι συνέπειες που πρέπει να εξανθούν. Αν τα γνωρίζουν και οι δύο, Μπορεί να υπάρχουν μειονεκτήματα, αλλά ε, όταν είναι από νωρίς η διαβούλευση θα τα δέχονται ε, όλοι. Βεβαίω ε, διαμαρτυρίε θα υπάρχουν, αυτή τη στιγμή ο πληθυσμό είναι σε άγνοια. Ευχαριστώ. Ποιο θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κανείς. Okay. The floor to you. Λοιπόν, από την αρχή, όταν έπαιρνα το λόγο για αυτή την έκθεση, ανέκαθεν υπογράμμιζα τη σπουδαιότητα του να υπάρχει ένας ε, οδηγός, ένα προηγούμενο σημαντικό σε αυτή μας την ε, αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Και όπως αποδείχθηκε η δουλειά που έγινε είναι πολύ σημαντική. Από πολλές απόψεις. Από τοπογραφική άποψη για πολλές τοπικές κοινότητες αλλά και από την άποψη των εργασιών ε, που πραγματοποιήθηκαν ε, στην ομάδα, στην επιτροπή μας, ε, στο πλαίσιο των συζητήσεων, όχι μόνο στο πλαίσιο των εργασιών στην Ελλάδα, των επισκέψεων σε διάφορες τοποθεσίες, που δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στο εξή. Όταν μια αντιπροσωπεία λάβει επαρκείς πληροφορίες ε, και σωστή καθοδήγηση σε μια τοποθεσία, όταν οι Έλληνες ευρωβουλευτές, και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα, ε, ε, επιδεικνύουν μεγάλη επιμέλεια διότι διαρκώς ήταν δίπλα μας ε, ακόμη και αν δεν ήταν οι ε, μέλη της αντιπροσωπείας μας βοήθησαν εξαιρετικά διότι ε, γνωρίζουν τα προβλήματα πολύ καλύτερα από τους βουλευτές των άλλων χωρών είναι φυσικό διότι έχουν επαφή με τα προβλήματα της Ελλάδας από την άλλη εγώ επέμεινα κοιτώντα ειδικότερα στο κέντρο της Πελοποννήσου προβλήματα που ναι είναι σημαντικά και σοβαρά όπως και σε άλλα μέρη αλλά υπάρχει και αυτό το θέμα του αμίαντου προβλήματα πολύ πιο δύσκολο να, για, να επιληθούν κυρίως και επειδή το υπέδαφος της Ελλάδας γεωλογικά περιλαμβάνει πολλές υδρολογικές δομές αόρατες αλλά και σε ένα μέρος ε, έτσι, σημαντικών γεωλογικών χαρακτηριστικών ε, μέσα στον χρόνο μπορεί να δημιουργηθούν ε, ακόμη σοβαρότερα προβλήματα. Η τροπολογία μου λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση υποδείκνυε. Για να συνοψίσω πρέπει να πω ότι αυτή η έκθεση αυτή τη δραστηριότητα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα κατά την απόψή μου και για πολλέ άλλες ενδεχομένω μελλοντικέ δραστηριότητες του ίδιου είδου, αλλά όχι μόνο αυτού του είδου. κατά την απόψή μου στην προηγούμενη περίπτωση δεν πρόκειται μόνο για τα αποτελέσματα που είναι ικανοποιητικά και οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν και σε άλλες δραστηριότητες, ίσως όχι για όλες, αλλά σε αρκετές. Πιστεύω διότι για να γίνεται σωστό σχεδιασμός, ε, ε, όταν γίνεται σωστό σχεδιασμός, ε, τα αποτελέσματα αργά ή γρήγορα είναι ικανοποιητικά, όπως συνέβη με αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δίνω τώρα το λόγο για τρία λεπτά στον ε, αναφερόμενο που είναι εδώ παρόν και που ζήτησε να παρέμβει για τρία λεπτά ε, στον κύριο Γκίκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι υποβουλευτέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και από πλευρά μου και από πλευρά των κατοίκων που ήρθατε. Είδατε το τι γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά με τους ε, υποκατασκευή χιτά και υπολειτουργία χιτά. Θεωρώ σημαντική την παρουσία μου στη συνεδρίαση αυτή όπως και σε άλλες συνεδριάσεις γιατί έτσι μας δίνεται η δυνατότητα με τον τρόπο αυτό να επικοινωνούμε με το κέντρο λήψης των αποφάσεων των επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα μας δίταξε δημοκρατία, πολιτισμό, αθλητισμό, φιλοσοφία, τέχνη. Φτιάξαμε Ακρόπολη, Παρθενώνα και άλλα πολλά. Δυστυχώς, εν έτη 2014 καταφέραμε ακόμα και ως κράτος, <clears throat> ως κράτος δεν καταφέραμε ακόμα ως κράτος να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας ή καλύτερα δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα να δούμε τα απορρίμματά μας ως προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε ανελαίτες απειλές από όλες τις ευρωπαϊκές επιτροπές και μας εκβιάζεται με τεράστια πρόστιμα για τους ανεκτέλετους χαδά. Αναρωτηθήκατε άραγε γιατί συμβαίνει αυτό. Γίνεται σωστή ανακύκλωση στην Ελλάδα. Εφαρμόζεται η οδηγία πλαίσιο 98-2008 Είστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις μας ως κράτος όσον αφορά την ανακύκλωση μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη στο θέμα της ανακύκλωσης μπαταριών. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να ανακυκλώσουμε. Μα φυσικά γιατί πολεμάνε την ανακύκλωση. Η σωστή ιεράρχηση είναι πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και στο τέλος έρχεται η διάθεση. Εμείς πάμε αντίθετα. Και αυτό γιατί έτσι συμφέρει τους εργολάβους, τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Η αναφορά Γκίκας Δαμάσκος που συζητάμε μαζί με την αναφορά του κ. Παπαδεγενόπουλου με 2.500 υπογραφές δεν έχει να κάνει μόνο με το γραμματικό, τουλάχιστον με τη δική μας αναφορά, καταγγέλνουμε όλο το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων πανελλαδικά. Στην περίπτωση του χιτά Φιλής, το μεγαλύτερο σκουπιδότοπο της Ευρώπης, δεν θα αναφερθώ σήμερα, έχω κάνει αναφορά, έχει πετύχει αριθμό, πετήτη 17-10-2013, και θα ήθελα την επόμενη φορά όταν θα συζητηθεί να είναι εδώ και ο κύριος Δαμάσκος ή Προσινάτ και κάτοικοι της περιοχής της φυλής και τότε να δούμε η Κομισιόν τι θα μας απαντήσει. Στην περίπτωση του γραμματικού, το έργο αυτό είναι ένα οικονομικό και οικολογικό σκάνδαλο. Τα μοναδικά κριτήρια για να κατασκευάσουν το έργο στο γραμματικό ήταν το λιγότερο πολιτικό κόστος και η λιγότερη πολιτική αντίδραση. Έτσι γίνονται τα έργα στην Ελλάδα. Έτσι κατασκευάζονται τα έργα. Το έργο αυτό είναι υπερδιαστολογισμένο, δεν προωθείται η ανακύκλωση αφού είναι μέρος της υλοποίησης του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, αλλά θέλει τα απορρίμματα να παραμένουν σύμμικτα. Την ώρα που ακόμα και η πρόσφατη έκθεση με αριθμό 20 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για το 2012 θέτει σε αμφισβήτηση τη χρηματοδότηση υποδομών επεξεργασίας σύμικτων απορριμμάτων. Έλεγχος που διεξήχθη σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία. Τι άλλο θέλετε να σας πούμε. Επίσης, στην περίπτωση του χιτά γραμματικού υπάρχουν πρόδειλα σφάλματα που η Κομισιόν μέχρι σήμερα αδυνατούσε να δει και εξακολουθεί να μην βλέπει. Το χειρότερο, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απέκρυψε και τα διερχόμενα ρέματα από την περιοχή κατασκευής του χιτά. Και πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος με το πάρτι και την κοροϊδία και το φαγοπότι που γίνεται μέχρι σήμερα με τις περιβαλλοντολικές μελέτες. Γιατί λοιπόν τους αφήνετε. Δώστε κίνητρα στους πολίτες <clears throat> και θα δείτε για πότε θα γίνει η ανακύκλωση και πότε θα σταματήσουν να ανεκτέλεστε στη χαδά. Με τον παρόσχεδιασμό, το μοναδικά κίνητρα <clears throat> που δίνεται είναι στους εργολάβους. Σας ζητάμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας, πόσο μάλιστα και μετά την επισκεψή σας, στον υποκατασκευή Χιτά, στους υποκατασκευείς χιτά που είδατε στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το γραμματικό. Παρακαλούμε θερμά όλους τους ευρωβουλευτές να δώσετε ένα τέλος σε όλο αυτό το οικονομικό και οικολογικό έγκλημα που συντελείται και στο γραμματικό και να, και να μην επιτρέψετε να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Είναι λίγος ο χρόνος που μου δίνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά και πάλι ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και σας δυστυχώς ε, είναι περιορισμένος ο χρόνος για όλους μας. Ε, θα θέλαμε όλοι να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτά τα ζητήματα που μας ε, παρουσιάζουν οι πολίτες. Ξαναδίνω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή, στον πρόεδρο της αντιπροσωπείας, τον συνάδελφο Τρουγκάης, για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω σημειώσει όλα τα σχόλια των συναδέλφων. Σημείωσα και όλες τις προτάσεις σας και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον μέχρι την τελική εκπόνηση του εγγράφου. Κυρία Πρόεδρε, θα τα συμπεριλάβουμε αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χουντή. Τα συμπεράσματα αυτά και οι προτάσεις του είναι πολύ χρήσιμα, γιατί όπως γνωρίζετε τα συμπεράσματα, κύριε Χούντι, είναι ανοιχτά. Μπορούν να βελτιωθούν, να συμπληρωθούν με τροπολογίες. Ε, εμείς ε, συμμετέχουμε στην εκπόνηση αυτού του εγγράφου όλοι μας. Και ο κύριος Μπαλτίνη είπε κάτι πολύ εύστοχο. Αυτό που έχει σημασία είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το ταξίδι και σε αυτό το έγγραφο. Μπορούμε βεβαίως να το συμπληρώσουμε με άλλες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για τη βελτίωση, όπως είπε και ο κύριος Μπαλτίνη, και βεβαίως εσείς θα συνεισφέρετε και σε εσά εναπόκειται ε, να κάνετε τις προτάσεις σας για το έγγραφο. Ο κύριος Αγκουράκης είπε, ναι είναι γεγονός ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου και εμείς θα θέλαμε να δούμε και άλλα προβλήματα. Και εσείς οι ίδιοι οι Έλληνες έχετε εντοπίσει προβλήματα, οι Έλληνες συνάδελφοι που δεν μπορούσαμε να δούμε εμείς όλες αυτές τις χωματερές και τα προβλήματα που υπάρχουν ε, ανά την επικράτεια στην Ελλάδα. Ε, είναι καλό να μας το επισημαίνετε. Το ξέρω ότι είναι η κορφή του Παγόβουνου και μόνο, αλλά κάναμε μια προσπάθεια. Έχουμε πείγνωση ότι δεν μπορέσαμε να τα δούμε όλα. Αλλά δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι για την Επιτροπή Αναφορών και για σας τους ίδιους στην ελληνική αντιπροσωπεία, ανεξαρτήτως κόμματος, ε, ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η αποστολή. Μου είπατε προηγουμένως το θέμα των κυρώσεων και τι σημασία έχει αυτό. Μα εμεί δικαστέ δεν είμαστε για να επιβάλλουμε κυρώσει. Το γνωρίζετε, δεν αποφαίνεται η Επιτροπή Αναφορών. Άλλοι λαμβάνουν τι αποφάσει για να πέσει η ράβδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, α πούμε, θα πρέπει να ρωτήσει τι γίνεται, να ρωτήσουμε και εμεί στην Επιτροπή πώ θα συνεχίσουν να αναλύουν την κατάσταση, πώ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν αυτέ τι εργασίε, τα κονδύλια που πηγαίνουν στην Ελλάδα για τέτοια θέματα. Ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, παρακαλώ να απευθύνουμε αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, θα είναι πιο ικανοποιημένοι οι πολίτες Τώρα εμείς η Επιτροπή Αναφορών θα προτείνουμε λύσεις στους πολίτες, να ζητήσουμε κυρώσεις. Ε, είναι ωραία αυτά επικοινωνιακά και για πηχαίους τίτλους ε, ζητάμε κυρώσεις, αλλά όπως γνωρίζει πολύ καλά ο αγαπητός ε, φίλος μου ο κύριος Αγκουράκης, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Εμείς είμαστε Επιτροπή Αναφορών, παρατηρούμε, καταγγέλουμε, συστάσεις απευθύνουμε, αλλά όχι κυρώσεις. Άλλοι έχουν αυτό το έργο στους ώμους τους. Για τον κύριο Σαλαβράκο. Είπε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συστάσεις 6-7-8. Το σημειώνω βεβαίως και θα το πράξουμε και παρακαλώ το φίλο μου κύριο Σαλαβράκο να μας βοηθήσει και εκείνο με προτάσεις. Γι' αυτό έχει ανοίξει προθεσμία για τις τροπολογίες για να μπορέσουμε και εμείς να βελτιώσουμε το κείμενο και τις συστάσεις που έχουμε υποβάλει. Έχετε το έγγραφο στα χέρια σας και παρακαλώ τις προτάσεις σας. Σημειώνω αυτά που είπατε θα προσπαθήσουμε και εμείς να βελτιώσουμε το κείμενο. Και τέλος κυρία Πρόεδρε, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όπως και στην αρχή όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την αποστολή και στην εκπόνηση του κειμένου. Και αναμφίβολα, επαναλαμβάνω, είμαι στη διάθεσή σας για να βελτιώσουμε το κείμενο μέχρι την τελική ψηφοφορία για να ψηφιστεί και να εγκριθεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε σένα Κάρλος για τη δουλειά σου. Εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους συναδέλφους όπως ακούσαμε. Η έκθεση αυτή θα εγκριθεί στην επόμενη συνόδο του Φεβρουαρίου κατά την οποία θα έχουμε και τη συμβολή των εθνικών αρχών. Πιστεύω σημαντική συμβολή αυτή για να ε, αρθούν οι περαιτέρω αμφιβολίες που έχουν προκύψει κατά την αποστολή και κατά τη συζήτηση των αναφορών. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο και Επαναρχόμαστε με τον συνάδελφο τον κύριο Σαλαβράκο στο σημείο 15 που είχαμε αναβάλει μέχρι να επανέλθει ο κύριο Συγητή. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Σαλαβράκο για την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να σα ευχαριστήσω σχετικά με τι τροπολογίε που καταθέσατε στην εκθεσή μου. Σα έχω αποστείλει το κείμενο με τι προτινόμενε συμβαστικέ τροπολογίε και περιμένω να ακούσω τα δικά σα σχόλια από αυτό και νομίζω ότι λόγω και της ε, σημαντικότητας του θέματος που αφορά την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα και το μέλλον τους, πρέπει να το δούμε όλοι και σε συνεργασία και με πολύ προσοχή. Εγώ είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε συζήτηση για την βελτίωση αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλαβράκο. Πριν αρχίσει η συζήτηση νομίζω θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. κυρία Στόκουελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σε ευχαριστήσω για το θέμα της Ιθαγένειας 2013 έκθεση και φυσικά θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πραγματικά η κατάλληλη στιγμή πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές να αναφερθούμε σε αυτό το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, αυτό βεβαίως ε, αφορά εξίσου και τα κράτη-μέλη αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων. Πολλά έχουν ήδη γίνει ιδιαίτερα μετά την έκθεση που αφορά το ίδιο θέμα του 2010 και αυτό φαίνεται και από τον ισότοπο Europa. 25 δράσεις αναλύθηκαν το 2010 και οι περισσότερες από αυτές έχουν ε, υλοποιηθεί πέρσι παραδείγματος χάρη το πακέτο για τα δικαιώματα των ε, ταξιδιωτών, των επιβατών και όσον αφορά την έκθεση για το 2013, κάποια έχουν ήδη υλοποιηθεί για τις ε, μικρές ε, διαμάχες παραδείγματο χάρη, το θέμα της κατάρτισης, γιούρες, εξυγχρονισμός του γιούρες που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και πριν τα Χριστούγεννα ξεκινήσαμε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα τη δυνατότητα διαμαρτυρίας και ανταλλαγής πληροφοριών των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Πολλά λοιπόν έχουν ήδη υλοποιηθεί, όχι όλα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και φυσικά εδώ χρειάζεται επιτάχυνση της διαδικασίας για το καλό και προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και ε, συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τις ε, επιπτώσεις της Ευρώπης για αυτούς, για τις οικογένειές τους και αυτό εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών. Χρειάζεται λοιπόν ενημέρωση, χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης και φυσικά ε, θεωρώ θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Αρχίζει λοιπόν ο ε, κατάλογος των ομιλητών. Πρώτος ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σημειώσω κάτι που έχω πει προσωπικά και στον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση, πολύ ισόρροπη και ε, περιλαμβάνει πολλά στοιχεία τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και με τον τρόπο που έχουν διατυπωθεί. Ε, να πω μόνο ότι εκτός από όλα αυτά υπάρχουν και κάποια σημεία για τα οποία νομίζω ότι χρειάζεται να συζητηθούν. Ευθύ εξ αρχή ε, θα ήθελα να απευθυνθώ στην εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συμφωνήσω ρητά και μαζί τη. Νομίζω ότι στην έκθεση ε, θα ήταν πάρα πολύ σκόπιμο να δούμε από τα 25 μέτρα που έχουν ε, εξαγγελθεί ε, ότι έχουν υλοποιηθεί κιόλα. Αυτό είναι ένα παράγον που δημιουργεί εμπιστοσύνη στα μάτια των πολιτών. Ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεκπεραιώνονται οι εργασίε και έχουν για αποτέλεσμα συγκεκριμένο και αυτό. Και είναι σημαντικό για μένα. Τώρα, για κάποια θέματα πολύ σύντομα θέλω να τα περιγράψω. Να σκεφτούμε πώς θα χειριστούμε με μονομένα σημεία όταν πρόκειται για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη που είναι ένα πολύτιμο επίτευγμα και κατάκτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες. Αυτό λοιπόν το θέμα δεν θέλω να το συνδέσω απολύτως με τα προβλήματα της πολιτικής λιτότητας. Ε, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να κάνουμε τέτοια σύνδεση και να ασχολούμαστε εκτενώς με τελείως διαφορετικά πράγματα από την ίδια την ιδιότητα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Ε, ας πούμε, υπάρχει το αίτημα επιθυμία για εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτό έρχεται σε κατάφορη αντίφαση με την επικουρικότητα, με την εθνική νομοθεσία. Δεν έχει νόημα τώρα να ζητάμε τον ουρανό με τα άστρα ε, και άσχετα πράγματα. Το ίδιο ισχύει ε, με τα δικαιώματα ε, υπηκών τρίτων χωρών. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν αλλού. Τι δουλειά έχει ε, η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πρόκειται ακριβώς για πολίτες της Ένωσης όχι τρίτων χωρών και κάποια άλλα θέματα που θα με ενδιαφέραν πάρα πολύ να διευκρινιστούν σε συνομιλίες μπορώ να ρωτήσω και με μονομένου συναδέλφου για να δω τι εννοούν, γιατί δεν έχω καταλάβει ε, όλα τα σημεία που ζητούν. Υπάρχουν κάποιε συμβαστικέ προτάσει που έχω επίση ερωτηματικά, γιατί εν μέρη. Βρίσκω τους συμβιβασμούς πάρα πολύ μακροσκελείς και θα ήθελα να μου εξηγηθεί ε, το θέμα. Ή άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με πρόσφυγες. Τι σχέση έχει αυτό με την ηθαγένεια. Αλλά παρακαλώ να μην θεωρηθεί αυτό αρνητική κριτική. Το αντίθετο, να τονίσω και πάλι ότι είναι εξαιρετική η έκθεση και βάση ε, στην οποία όμως θα ήθελα να διευκρινιστούν πολλά θέματα για να γίνει τέλεια η έκθεση. Ο Σκιώδης εισηγητής Έχω αυτή τη φιλοδοξία, δεν το κρύβω και γι' αυτό σας ζητώ να ληφθούν υπόψη ορισμένα σημεία. Ότι χρειάζεται μια μικρή συνεδρία των σκιωδών, αλλά αυτό θα τα πω διμερώς με τον εισηγητή και άτυπα θα το λύσουμε. Ευχαριστώ και τη γραμματεία βεβαίως για τη συνεισφορά ε, για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέκερ. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και κατά την πρώτη συζήτηση της έκθεσης του συναδέλφου του Σαλαβράκου αλλά και τώρα που συζητάμε τις τροπολογίες θέλω να επαναλάβω ότι ο συνάδελφος έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και πολύ εμπεριστατωμένη σε ένα θέμα που όπως αποδείχθηκε και από την προηγούμενη ομιλία χρειάζεται πολύ προσεκτική, πολύ υπεύθυνη, πολύ δημοκρατική ευαισθησία για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Ε, κύριε Πρόεδρε, έχω καταθέσει τροπολογίες όπως και η κυρία Βερζιά εκ μέρους της ΓΚΟΕ και ο καθένας ξεχωριστά τροπολογίες ε, τις οποίες προφανώς έχει πάρει υπόψη ο κύριος Σαλαβράκος. Ορισμένες από αυτές έχουν ενσωματωθεί κάποιες άλλες δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμηση του, του εισηγητή για να δούμε και την τελική μας στάση σε σχέση με τις συμβιβαστικές προτάσεις, για να είμαι σύντομος, συμβιβαστικές τροπολογίες, ε, είμαστε σύμφωνοι, είμαι σύμφωνος, στις τροπολογίες, τις συμβιβαστικές επαναλαμβάνω, με τον αριθμό 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Δεν λέω σε τι αναφέρεται, γιατί δεν έχουμε ίσως χρόνο, αλλά έτσι όπως συμπυκνώνει τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σε συμβιβαστικέ τροπολογίες κατά βάση μας βρίσκουν σύμφωνος. Οι ενστάσεις μου ή τα ερωτηματικά μου είναι στις πρώτες δύο συμβιβαστικές προτάσεις. Και πιο αναλυτικά, σε σχέση με την πρώτη συμβιβαστική πρόταση, στο βαθμό που περιλαμβάνει τροπολογία που αναφέρει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυση τις οικονομικές ελευθερίες των πολιτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν συμφωνώ με αυτή τη διατύπωση, αλλά αν θέλετε δεν είναι θέμα να το διατυπώσουμε, δεν συμφωνούν τα γεγονότα. Τα γεγονότα που ζούμε αυτή την περίοδο με τον έναν τον άλλο τρόπο, η κρίση γενικώ στην Ευρώπη και σε ορισμένε ιδιαίτερα χώρε, δεν νομίζω ότι χωράει δεύτερη γνώμη ότι τουλάχιστον στον τομέα των οικονομικών ελευθεριών δικαιωμάτων κατ' επέκταση των πολιτών, η συνθήκη της Λισαβόνας τα κατοχυρώνει. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα της παρατήρησης, διότι αντιστρέφει τα γεγονότα, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και η ίδια παρατήρηση σχετικά με το πόση εγγύηση και πόση εμπιστοσύνη μπορεί να έχει ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ψήφιση και την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρεται και στη συμβαστική 2 και ιδιαίτερα στην τροπολογία 86. Για αυτούς τους λόγους, για αυτό το λόγο, στις δύο συμβιβαστικές έχω ερωτηματικά αν ε, δεν, δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Με αυτή την έννοια. Τέλος θέλω να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που δεν περιλαμβάνουν τις συμβιβαστικές και που έχουν κατατεθεί και τις θεωρώ σημαντικές. Η μία τροπολογία κύριε Πρόεδρε είναι η τροπολογία 60 στην οποία νομίζω και ο κύριος Αλαβράκος το γνωρίζει πολύ καλά ως Έλλην ότι θα πρέπει να δίδεται το δικαίωμα στους πολίτες μιας χώρας να μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές της χώρας καταγωγής από τη χώρα που ζουν. Δηλαδή να σας το πω πιο απλά, ενδεχομένως οι Έλληνες πολίτες να είναι οι μόνοι πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν τη δυνατότητα από την χώρα που μένουν διαμονής να ψηφίσουν για τις εκλογές της χώρας τους, για τις εθνικές εκλογές. Αυτό πρέπει να επισημαίνεται, αυτό πρέπει να διεκδικείται, αυτό πρέπει να σημειώνεται πολύ περισσότερο μάλιστα που λόγω της κρίσης έχουμε νέα μεταναστευτικά ρεύματα από την Ελλάδα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες που δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν για οικονομικούς λόγους και να έρθουν να ψηφίσουν, να μπορούν να ψηφίσουν στη χώρα που κατοικούν πια και δουλεύουν και που έχουν δικαίωμα να ασκήσουν πολιτικά Την πολιτικά τους δικαιώματα, συγγνώμη. Τέλος αναφέρομαι στην τροπολογία 35 Έχουμε καταθέσει με την κυρία Βερζέα την τροπολογία ότι είναι απαράδεκτο, θεωρούμε απαράδεκτο, το γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει θυγεί και άλλες φορές, ότι στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού και της προσοχής στρέφεται στο πρόγραμμα Μνήμη. Εκεί επιχειρείται να διαδοθεί η αντίληψη και να μάλιστα και να διδαχθεί η αντίληψη ότι ο ναζισμός είναι, εξομοιώνεται με τον κομμουνισμό. Δεν το αντιμετωπίζω μόνο από ιδεολογική αφετηρία το θέμα. Μια τέτοια προσπάθεια αγαπητοί συνάδελφοι είναι παραχάραξη της ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας της Ευρώπης και αν ο Ευρωπαίος πολίτης δεν γνωρίζει καλά την ιστορία καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να σκίσει αντίστοιχα τα δικαιώματα επομένως έχει άμεση πολιτική σκοπιμότητα αυτό που γίνεται. Το δεύτερο είναι επικίνδυνο ένα τέτοιο πράγμα και πρέπει, είναι επικίνδυνο και από την άποψη της γνωριμίας του ενός λαού και του άλλου που μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βρέθηκε ο ένας δίπλα των άλλον, είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, όπου συναντιούνται ιστορίες και πολιτισμοί και επομένως τέτοιες αντιλήψεις δεν βοηθάνε για να μπορέσει να διαμορφωθεί η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη και κατά, και κατά βάση να διεκδικηθεί η ηθαγένεια ή και τι σημαίνει η ηθαγένεια και με αυτή την έννοια θα ήθελα να, σας, να δώσετε την δέουσα προσοχή, αγαπητοί συνάδελφοι, για αυτούς τους λόγους. Ε, επαναλαμβάνω, στις ε, ε, έξι από τις οκτώ συμβιβαστικές συμφωνούμε, στις δύο υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις και από τις τροπολογίες που κατέθεσα ήθελα να υπογραμμίσω τις δύο αυτές περιπτώσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χοντή. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Στανόκα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι περίεργο θέμα η ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ε, την περασμένη εβδομάδα κατά τη Σύνοδο συζητήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και όταν εξήγησα εγώ με τη δήλωσή μου την ε, αποχή μου για αυτό το ψήφισμα μου είπαν ότι δεν υπάρχει διότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγενή είναι είναι απλά ένα παράγωγο της εθνικής ε, υπηκότητας δεν υπάρχει κανένας που να έχει υπηκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να μην έχει υπηκότητα ενός κράτους μέλους. Αυτή είναι η διχογνωμία εδώ στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την, ελληνική, την ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Θα πρέπει όμως να έχει κάποια προστιθέμενη αξία είτε να λειτουργεί ως έχει ή να αποτελεί απλό παράγωγο τη ηθαγένειας ενός κράτους μέλους. Εγώ είμαι υπέρ της πρώτης προσέγγισης. Τον, ε, έχει μεγαλύτερη αξία η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το να χορηγείται η ηθαγένεια αυτή σε μια σειρά ατόμων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχουν την ηθαγένεια οποιοδήποτε κράτους μέλους και πρώτη υποψήφοι για μια τέτοια ηθαγένεια θα ήταν ε, οι επωνομαζόμενοι μη πολίτες ε, της Λετωνίας και της Εσθονίας ε, των οποίων τη διαβατήρια εκδόθηκαν ε, καλυπτόμενοι από τη διπλωματική προστασία αλλά χωρίς πλήρη δικαιώματα στα κράτη-μέλη αυτά. Αναφορές για αυτά τα θέματα έχουν υποβληθεί από τη Λετωνία και την Εστονία. Δεν ήταν το 2013 βέβαια, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Και τα εν λόγω άτομα δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα ψήφου ε, ή το να είναι υποψήφιοι σε εκλογές κτλ. Η τροπολογία μου που αφορά αυτό το πρόβλημα δεν συμπεριληφθήκε στη Συμβαστική έπτα που καλύπτει μόνο τα προβλήματα των ευρωεκλογών. Συμφωνώ με τη δήλωση με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμβιβαστική. Και σε μία από τις δικές μου τροπολογίες ε, θέτουμε το θέμα της ε, μικρής συμμετοχής των πολιτών ε, ενός κράτους μέλους που διαμένουν σε ένα άλλο κράτος μέλος στις ε, ευρωεκλογέ ε, λοιπόν, η τις κοινοβουλευτικέ εκλογες του λογω κρατους μελους εμενα ειναι ταλο υποψηφιο λυπουμε λοιπον που αυτη η ιδεα του να παρέχουμε ε, σε μόνιμου κατοίκου το δικαίωμα να συμμετέχουν στι εκλογέ, αποτελεί πρακτική σε ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Μισά μισά είναι χωρισμένα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη χορήγηση αυτού του δικαιώματο, των εκλογικών δικαιωμάτων, ενεργών εκλογικών δικαιωμάτων σε μόνιμου κατοίκου που δεν είναι πολίτε, δεν έχουν την υπηκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκ μέρου αυτών ε, μιλάω εγώ κάνοντα αυτέ τι προτάσει. Βλέπετε όταν η Μάλτα χορηγεί ηθαγένεια σε ξένους ε, τότε ευαισθητοποιούμαστε και λέμε ότι είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα αλλά όταν τίθε το ζήτημα των απάτριδων που έχουν γεννηθεί στα κράτη-μέλη τότε μας λέει η Κομισιόν ότι δεν είναι ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό και ότι αποτελεί αρμοδιότητα του κρατούς μέλους. Δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν χρησιμοποιούνται όσον αφορά αυτή τη ε, διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών όσον αφορά την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πιστεύω είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που τίθεται, το οποίο δεν έχει επιληθεί και που τέθηκε από την Επιτροπή μας. Είχαμε μία έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ε, και συμμετείχα και εγώ και οι δικές μου προτάσεις ε, αναφέρονταν στο ζήτημα αλλά δεν είχαν υποστήριξη από τη δεξιά ε, ομάδα του Κοινοβουλίου. Σκοπό ήταν να δοθεί προστιθέμενη αξία στην ηθαγένεια. Είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί σωστά. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Σδενόκα. Ο κύριος Μποστινάρο έχει το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν uh, στηρίζουμε αυτή την uh, έκθεση, το σχέδιο έκθεσης, καθώς και το γεγονός ότι ο κύριος Αλαβράκος κατάφερε να ενσωματώσει στις συμβαστικές προτάσεις της προτάσεις των σκιωδών ε, και εδώ αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα στις δικές μου προτάσεις με η εισηγητής ε, των ε, σοσιαλιστών και δημοκρατών. Πιστεύω πραγματικά ότι οι σκέψεις της κυρίας Τάνοκα είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Όντως υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν ούτε καν στην ε, κατηγορία των ε, πολιτών δευτέρας κατηγορίας. Δηλαδή πρόκειται για άτομα που έχουν γεννηθεί στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές υπάρχει δικαστική απόφαση που τους στερεί αυτό το πολύ συγκεκριμένο συνταγματικό τους δικαίωμα και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρούμε μια λύση. Στις συζητήσεις μας λοιπόν με τους κοιόδης συζητητές θα πρέπει να βρεθεί μια διατύπωση σαφής που να αντικατοπτρίζει αυτό το θέμα και να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σύντομα στο μέλλον να βρει λύση, να βρει ένα τρόπο να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Την ίδια ώρα θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να ενισχύσουμε και να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν όλα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, ακόμα και των Ρουμάνων, ακόμα και των ε, Βουλγάρων. Πολλές φορές βλέπουμε αυτοί οι πολίτες να προσδιορίζονται με έναν απαράδεκτο τρόπο. Δηλαδή σε λίγο θα τη ζητήσουμε να έχουμε ναι, και κάποια ενδεικτικά στοιχεία όπως το κίτρινο αστέρι που είχαν οι Εβραίοι στον πόλεμο. Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει πραγματικά να στείλουμε ένα μήνυμα. Η Επιτροπή των Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στέλνει ένα σαφέστατο μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε δύο κατηγορίες Ευρωπαίων πολιτών, πρώτης και δεύτερες κατηγορίες. όλοι όσοι γεννήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Γι' αυτό ακριβώς και πιστεύω ότι αυτές οι ιδέες θα πρέπει να μπουν με έντονο τρόπο και να τις υπογραμμίσουμε στην έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή γιατί έχει δείξει πολύ ανοιχτό πνεύμα και πιστεύω ότι θα βρεθούν λύσεις και για όλα αυτά τα πολιτικά θέματα. Πρόκειται για μένα για το DNA της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουστινάρου. Το λόγο έχει για να κλείσει ο εισηγητής μας ο κύριος Αλαβράκος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν πάνω στην έκθεση ε, θεωρώ την έκθεση όλων μας και, με αυτό το σκεπτικό και την προηγούμενη φορά που αναφέρθηκα στην έκθεση αλλά και τώρα θα μιλήσω. Έχουμε ένα θέμα και πρέπει να αναπτύξουμε το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα αυτό νόμικα ο ηθαγένεια Ευρωπαίο πολίτη όπως το τόνισε και η κυρία Σντάνοκα είναι παράγωγο. Δεν μπορούμε να μεταβάλουμε την νομική μορφή του θέματος με τον οποίο ασχολούμαστε τώρα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να περάσουμε μέσα ιδέες που θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό συμβόλαιο ε, όπως κάποτε που νεότεροι είχαμε την έμπνευση από το Ρουσό και από τον Μοντεσκέ, ναι. αλλά νομικό κείμενο το οποίο θα μπει σε περιπτωσιολογία και δεν θα είναι κείμενο γενικών αρχών δεν μπορεί να υπάρξει και δεν μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα διότι θα τύχει των αντιδράσεων των κρατών μελών. Για να έχουμε ένα αποτέλεσμα από αυτή την έκθεση και μια ουσία από αυτή την έκθεση θα πρέπει κατά την άποψή μου να δώσουμε βασικές γενικές αρχές οι οποίες δεν προκαλούν την αρχή της επικουρικότητας διότι όπως ξέρετε ε, κατά το γέννη έχω, δηλαδή σήμερα που μιλάμε, οι τάσεις μέσα στην Ευρώπη είναι και η αντίδραση μέσα στην Ευρώπη είναι ο περιορισμός από τη μια πλευρά των, από, τους ε, της εθνικής κυριαρχίας των κρατών με τη δημιουργία της πολιτικής ενώσεως και από την άλλη πλευρά η αντίδραση η οποία λέει ότι όχι να μειώσουμε την Ευρώπη και να αυξήσουμε την ε, εθνική κυριαρχία. Με την έκθεση μου αυτή προσπάθησα να κινηθώ στο μέσον συμβιβαστικά πάνω στις υπάρχουσες τάσεις αυτή την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τις οποίες θα τις δούμε και στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ε, με τον κύριο Μπέκερ είχαμε πάντα καλή συνεργασία και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την καλή συνεργασία να βρούμε τον τρόπο ε, ενσωματώσεις αυτών των οποίων ε, θέλει. Με τον κύριο Χουντή έχουμε πρωτίστως καλή φιλία και τον ευχαριστώ που αποδέχεται αυτές τις ε, ε, ε συμβιβαστικές προτάσεις τις οποίες θα τον Στη συμβιβαστική 1 και 2 που αφορά την τροπολογία 60 και την τροπολογία 35. Η τροπολογία 35 Συμφωνώ μαζί του στο εξή, ότι δεν μπορώ να αξιομοιώσω τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. Βεβαίω. Αλλά δεν έχει θέση αυτή η τροπολογία, διότι προορίζεται για το κεφάλαιο μνήμη το οποίο δεν έχει γραφτεί. Δεν μπορώ επομένως σε γραπτό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προκαταλάβω το τι θα λέει αυτό το κεφάλαιο. Και νομίζω ότι ε, δεν ξέρω αν κάποιο γνωρίζει τι λέει. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει γραφεί ακόμη. Απλώ γράφεται ακόμη. Ε, γράφεται, δεν έχει, δεν έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή του. Επομένω νομίζω ότι θα κάνει κακό ακόμη και στι επιδιώξει του κυρίου Χουντή να έρθουμε προθύστερα να δώσουμε κατεύθυνση και να αναγνωρίσουμε τέτοιου είδου πράγματα ή διάφορα μυαλά τα οποία είναι νοσηρά να τα κατευθύνουμε προς τέτοιου είδους κατευθύνσεις. Στο 60 να δω και το είναι μισό λεπτό. Στο 60. Στο ε, έρχεται στο θέμα των εκλογικών δικαιωμάτων για τους υπηκόους των κρατών μελών. Υποτίθεται ότι η νομοθεσία εκλογής στα κράτη-μέλη και το βλέπουμε σε όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις ευρωπαϊκές εκλογές αφήνουν τις λεπτομέρειες στη βάση της αρχής της επικουρικότητας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι άλλοι ευρωβουλευτές έχουν εκλεγεί με ψήφο και άλλοι έχουν εκλεγεί με λίστα. Είναι ανάλογα με το τι συμβαίνει και τι αποδέχεται η κάθε χώρα στην νομοθεσία της. Δεν μπορεί επομένως να γίνει παρέμβαση κατά την άποψή μου η οποία να επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να ασκούν οι πολίτε το δικαίωμα ψήφου στι εθνικέ εκλογέ τη χώρα προελευσή του από το κράτο μέλο στο οποίο διαμένουν. Στην πράξη, όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή στι πρεσβείε του στο εξωτερικό το έχουν λύσει αυτό το θέμα πρακτικά. Διότι πηγαίνουν εκεί οι πολίτε κάτοικοι, πηγαίνουν στι πρεσβείε οι πολίτε κάτοικοι μια άλλη χώρα και ψηφίζουν. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα σε όλες τις πρεσβείες λειτουργεί η κάλπη. Έρχομαι τώρα στο θέμα της ε, κυρίας Σδάνοκα. Ε, Συμμερίζομαι τις απόψεις Δεν είναι παράλογες οι απόψεις. Ε, όλοι μιλάμε σε ένα πλαίσιο λογικής. Μάλιστα εμένα στην Ελλάδα ε, με κατακρίνουν πολιτικά διότι έχω πει ότι πλέον οι ιδεολογίες είναι για να τις συζητάμε με ουίσκι το βράδυ μετά τις 12 νομίζω ότι οι ιδεολογίες απλούστατα κατευθύνει κάθε ένα σε την ιδεολογία του που είναι σεβαστή και η ιδεολογία κατευθύνει σε έναν τρόπο επιλύσεως των προβλημάτων. Στον ίδιο τρόπο κατευθύνει και η λογική. Και νομίζω ότι λαγικά όλοι μιλάμε εδώ και άκουσα όλους τους συνεργάτες και, όλου όλους τους συναδέλφους οι οποίοι μίλησαν ε, πάρα πολύ λογικά. Ε, συνεπώς δεν μπορώ να θέσω ότι οι προτάσεις οι οποίες μου γίνονται για την τροποποίηση είναι ε, προτάσεις οι οποίες προεχόντως βασίζονται σε πολιτική ιδεολογία. Θεωρώ την κοινή λογική ότι μπορεί να κυριαρχήσει. Είδατε και το επισημάνατε κυρία Σντάνοκα το θέμα της Μάλτας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ωραίο να μιλάμε ο ένας άνθρωπος για τον άλλον και έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να μαλακώσουν τα ήθη. Άλλωστε, ξέρετε, ο ελληνικός πολιτισμός ε, θεωρεί ότι πάντων μέτρων είναι ο άνθρωπος. Βεβαίως οι Ρωμαίοι λένε ότι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος. Homo hominis lupus. Δηλαδή πρέπει να και εκεί να βρούμε κάποιο τη μέση. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να πω ότι θα συζητήσουμε το οτιδήποτε, είμαι ανοιχτό να συζητήσουμε το οτιδήποτε, αρκεί να εναρμονίζεται με την έκθεση και να, έχει, να κάνει την έκθεση αποτελεσματική. Να έχει κάποιο αποτέλεσμα την έκθεση. Εδώ δεν θέλω να επιχεί αυτή η έκθεση τις πολιτικές εντό εισαγωγικών για μένα απόψεις του καθενός μας. Πρέπει να απηχεί τη λογική του καθενός μας. Και όλοι μας έχουμε λογική. Και αναγνωρίζω στο φίλο μου τον κύριο Παστινάου πολύ λογική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλαβράκο. Συμφωνώ και εγώ με τα συγχαρητήρια των συναδέλφων. Όλες οι πολιτικές ομάδες σας συνεχάρισαν. Στα χέρια σας τώρα είναι η προσπάθεια ε, όσο μπορείτε να συντονίσετε τις διάφορες απόψεις. Το Φεβρουάριο θα ψηφίσουμε και ελπίζω και το λέω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έκκληση το μόνιμο πάγιο ε, δίκαιο αίτημα της κυρίας Δανόκα σε όλες τις συζητήσεις σε σχέση με αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες που είναι στο πουθενά μετέωροι άνθρωποι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βρούμε μια οριστική λύση για αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά και περνάμε αμέσως στο σημείο 18 αναφορά 1175 κάθετος 2012 της Τάνιας Τζάξον, Βρετανικής Ιθαγένειας, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο πυρηνικών αντιδραστήρων στο Hinkley Point, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απουσιάζει η συντάκτρια της αναφοράς. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Δον Σαντιάγο Μαρτίνεθ Ιγκλέσιας από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Όσον αφορά αυτή την αναφορά, η Επιτροπή γνωρίζει τους κινδύνους που έχει τα διάφορα και έχουμε ορίσει τα πρότυπα όσον αφορά τους κινδύνους που προκύπτουν από την κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων σε διεθνές επίπεδο ε, προτείνεται να περιορίζεται η ακτινοβολία από όλε τι ε, πρακτικέ ε, σε συγκεκριμένα όρια, τα σημερινά πρότυπα ασφαλεία ε, στην Ευρώπη. Προβλέπονται τα ίδια όρια του ενός μιλισίβερ το χρόνο. Η νέα οδηγία του Συμβουλίου για τα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας από την ακτινοβολία που υιοθετήθηκε 5 Δεκεμβρίου του 2013 επιβεβαιώνει την εγκυρότητα αυτών των ορίων και της προσέγγισης στις διαφορές ε, ηλικίες και φύλου. Όσον αφορά την κατασκευή των δύο πυρηνικών αντιδραστήρων ε, στο Hinkley Point, η Κομισιόν ε, έδωσε την αποψή της στη γνωμοδότηση της 12 Ιουλίου 2012 όπου βάσει με την προηγούμενη αξιολόγηση και τις συζητήσεις με τον επενδυτή η επένδυση εκπληρώνει τους στόχους της συνθήκης Ευρατών. Αποτελεί εθνική ευθύνη πρωταρχικά και αποτελεί ευθύνη του επενδυτή να εξασφαλίσει και του Εθνικού Ελεγκτικού Οργανισμού να ε, επαληθεύσει ότι τηρούνται τα όρια ασφαλείας ε, και ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμπεραντά των ε, stress test που έγινε στην Ευρώπη μετά από το ατύχημα στη Φουκουσίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τέιλορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις αυτές. Διάβασα την αναφορά και θεωρώ ότι η Κομισιόν δεν έχει εμβαθύνει επαρκώς ε, την εξέταση των ισχυρισμών ε, που περιλαμβάνονται στην αναφορά. Πιο συγκεκριμένα η αναφορά ε, αναφέρει ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν ασθενείες λόγω ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριμένα ο αναφερόμενος, η αναφερόμενη συσχετίζει την ακτινοβολία με κάποια ε, βλάβη στη γέννηση κοριτσιών. Επίσης αναφέρεται σε μια ε, έκθεση σχετική. Λέει λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες σε ασθενείς λόγω και ισχυρίζεται ότι και λέει, εδώ ότι ανησυχεί ότι οι άνθρωποι που ορίζουν τα πρότυπα ε, της ακτινοβολίας στην πλειοψηφία τους είναι άντρες. Πιστεύει λοιπόν ότι οι γυναίκες έχουν κάπως εκτοπιστεί από, αποκλειστεί από τις μελέτες αυτές. Πραγματικά λοιπόν θεωρώ ότι η Κομισιόν δεν έχει απαντήσει στην αναφορά με τρόπο ολοκληρωμένο όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις για τα διαφορετικά φύλλα ε, από ακτινοβολία χαμηλού επίπεδου. Υπάρχει τεράστια ποικιλία μελετών, ε, ειδικότερα μετά από τη Φουκουσίμα. Θα ήθελα λοιπόν περαιτέρω αιτιολόγηση της απάντησης αυτής προς την αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο το λόγο από τους συναδέλφους. Όχι. Μετά από τις δύο τοποθετήσεις συμπεραίνουμε ότι αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά για να δοθεί συνέχεια σε αυτό το θέμα. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 19. Είναι η αναφορά του κυρίου Πέταρ Τρογιάνσκι Βουλγαρική ηθαγένειας εξ ονόματος Ένωσης Άννα για την ελευθερία του λόγου σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες όσον αφορά πυρηνικούς σταθμούς στη Βουλγαρία. Αποουσιάζει ο αναφέρον, οπότε θα δώσουμε μέσα το λόγο ε, στον Σαντιάγο Μαρτίνης Εγκλέσης, Ξενόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την αναφορά αυτή, η πυρηνική ασφάλεια παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες ε, της Ευρατόμ του Συμβουλίου δίνονται ε, στα άρθρα 4 και 5 στις εθνικές αρχές. Ε, και ε, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή ε, της Βουλγαρίας θα πρέπει να διερευνήσει τα όσα λέγει η αναφορά και θα πρέπει η Βουλγαρία να αποφασίσει εάν θα χτιστεί ή όχι νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Ε, το επενδυτικό ε, άρθρο, σχέδιο συγγνώμη, θα πρέπει βάσει του άρθρου 41 να υποβληθεί. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή υιοθέτησε το 2008 την άποψη ότι όλες οι πτυχές σε λόγω επένδυσης ήταν σύμφωνες με τους στόχους της συνθήκης Ευρατόμ σε σχέση με το Κοσλοντούι και το μελλοντικό σταθμό και την υπερπαραγωγή ενέργειας σε σχέση με τις ανάγκες δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό να σχολιάσει. Είναι εθνική αρμοδιότητα. Δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σχολιάζει ζητήματα ποινικού δικαίου των κρατών μελών. Είναι αμυγός εθνική αρμοδιότητα, αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλει το λόγο από αυτού. Παρακαλώ. Ο κύριος Ιρασάμπαλ Μπέιτια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προφανώς έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ουσίας για τις αρμοδιότητες κτλ. Μια μικρή παρατήρηση. Τελευταία η πυρηνική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει νέα όθηση προωθείται μία ενέργεια που είναι πανάκριβη και άκρος επικίνδυνη και πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, όπως είδαμε στη Φουκουσίμα πριν από λίγα χρόνια. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μπει σε τέτοια θέματα ποινικού δικαίου ε, ως προς την αναφορά αυτή. Ούτε πρέπει να βασίσει τη γνώμη της στα ε, στοιχεία που μας δίνουν βουλγαρικές αρχές. Γιατί από ό,τι φαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά φαινομενικά τηρούν ε, τις ε, προδιαγραφές της Ένωσης. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, απλώς για μια άλλη φορά να διατρανώσω την αντίθεσή μας ε, προς την πυρηνική ενέργεια. Γιατί έχει ξανασηκώσει κεφάλι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέιτια για την τοποθέτησή σας αυτή. Άλλος ουδής Οπότε θα περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο 20 αναφορά 1666 κάθετος 2013 από ένα Ρουμάνο υπήκο, ρόταφλεδο εδώ. Α, ε, η προηγούμενη μένει ανοιχτή ή κλειστή, δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα να μείνει ανοιχτή η αφορά αυτή έτσι για πάνε για καλό και για κακό, συμφωνείτε. Ωραία, παραμένει ανοιχτή. Περνάμε στο σημείο 20, η αναφορά όπως σας έλεγα του κυρίου Πίταφ αρχικά. Ρουμανικής Ιθαγένειας, εξ ονόματος του συλλόγου, ώστε τις γειτονιές Νταμαροάγια και ε, το, το Βουκουρέστι μας. Σχετικά με την καζόμενη παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση μεγάλου αριθμού κτηρίου στην ιστορική περιοχή Παρσελάρια Μπασιλέσκου στο Βουκουρέστι. Είναι ο κύριος Πέτρο Τρούτα παρόν, ο ΠΙΤΑΦ. Και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Λέγομαι Πέτρου Τρούτσα και είμαι πρόεδρος αυτού του συλλόγου που δημιουργήθηκε επί τούτου για να σας ενημερώσουμε ότι δεν πρόκειται εδώ για καμία πολιτική τοποθέτηση κυρίες και κύριοι όπως παρουσίασα και στο παρελθόν ο σύλλογός μας για να σώσουμε την ε, συνοικία Δωμαράια και το Βουκουρέστι Νόη αναφέρεται στα διαμερίσματα του Βουκοριστίου. Υπάρχουν έξι με πολλές συνοικίες. Εμείς λοιπόν ουσιαστικά θέλουμε να αντιδράσουμε στις τοπικές αρχές, στην κοινότητα και στο Δήμο που θέλουν να καταστρέψουν τις συνοικίες μας παραβιάζοντας όλους τους νόμους που αφορούν την πολεοδομία, τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για δύο συνοικίες, Μπαζιλέσκο, που από το 1906 είναι διατηρητές περιοχές και φυσικά βρίσκονται και τις ιστορικές ε, συνοικίες από το 2004 της πόλης του Βουκουρεστίου. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα κτίρια τα οποία δεν πρέπει να πειραχτούν καθώς και πολύ συγκεκριμένες ε, επιφάνειες που πρέπει να παραμείνουν μη οικοδομήσιμες ε, καθώς και το πράσινο το οποίο καθορίζεται. Πρόκειται όμως εδώ για ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει την ε, οικοδόμηση κτηρίων χωρίς χώρους στάθμευση και χωρίς καμία πρόβλεψη για φύτευση δέντρων και επιφάνειες που θα πρέπει να παραμείνουν πράσινες. Πολλές φορές βλέπουμε μάλιστα παμπάλια δέντρα τα οποία θα εξαφανιστούν και βεβαίως μετά από την σύσταση του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι περιοχές αυτές πρέπει να παραμείνουν διατηρητές. Σήμερα όμως έχουν οικοδομηθεί παράνομα κτίρια, αυθαίρετα κτίρια που αρχικά δεν έπρεπε να ξεπερνούν τους δύο ορόφους. Σήμερα βλέπουμε στη θέση αυτών των κτιρίων καθώς και τις άδειες της πολεοδομίας να έχουν παραβιαστεί. Πρόκειται για παράνομη οικοδόμηση κτηρίων και κανείς ποτέ δεν προσέφυγε κατά αυτών οι οποίοι παραβίασαν την νομοθεσία. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για συνοικίες ε, της ε, πρωτεύουσα μας, οι οποίες ήταν και θα έπρεπε να παραμείνουν διατηρητές με μεγάλες πράσινες επιφάνειες. Σήμερα όμως βλέπουμε μεγάλα σύγχρονα κτίρια, πολυόροφα, τα οποία καταστρέφουν το περιβάλλον. Γι' αυτό και σας ζητούμε να λάβετε υπόψη σας ότι δεν πρόκειται για ένα τοπικό φαινόμενο. Υπάρχει παρόμοια ε, παράνομη οικοδόμηση κτηρίων και σε άλλες περιοχές. Και σήμερα βλέπουμε ότι ο έλεγχος από μέρους της ε, κυβέρνησης, των κεντρικών αρχών, είτε του Δήμου του Βουκουρεστίου, δεν έχουν απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στις αρμόδιες αρχές. Το μόνο που μας μένει αυτή τη στιγμή είναι να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη. Έχουμε απευθυνθεί και στον Δήμαρχο του διαμερίσματος αλλά και στον Δήμο της πόλης. 18 υποθέσεις εκκρεμούν μπροστά στην ρουμανική δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω πρόκειται για παράνομες διαδικασίες. Ξέρουμε όμως ότι αυτές οι διαδικασίες δυστυχώς παίρνουν χρόνο. Τρία με πέντε χρόνια μέχρι να έχουμε μια απόφαση. Γι' αυτό και σας ζητούμε να μας στηρίξετε, να μας βοηθήσετε και να προστατεύσετε τους Ρουμάνους πολίτες Και πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για δύο συνοικίες. Εγώ έχω γεννηθεί στην συνοικία, σε μια από αυτές τις δύο συνοικίες και πολύ θα θέλαμε να υπάρξουν περισσότερα λουλούδια, περισσότερη κήπη, περισσότερο πράσινο. Οι τοπικές αρχές βεβαίως αγνοούν την ε, επιθυμία των κατοίκων και αυτό βεβαίως μπορεί να οδηγήσει σε βίες συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων αυτών των περιοχών και αυτών που συνεχίζουν να οικοδομούν παράνομα. Σας ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρούτα. Πριν αρχίσει η συζήτηση θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Ντανιέλα Βαλέρη Αντρέη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά υποβλήθη πρόσφατα. Η Κομισιόν λοιπόν ακόμη αξιολογεί ποια από τις περιβαλλοντικές απαιτήσει εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή και τι έχει επιτευχθεί. Θα, σταλ, σταλεί το σχετικό έγγραφο. Ο κύριος Μποστινάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μέχρι εδώ τα ισπανικά μου. Πήγα λίγο στη Μάλαγα και έχω μάθει να λέω ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο και τους αναφέροντες. Πρόκειται κατά τύχη για την συνοικία στην οποία μένω στο Βουκουρέστι. Πρόκειται όμως για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι συνάδελφοι από την Ισπανία θα μου έλεγαν ότι τέτοιου είδους περιπτώσεις πρόκειται για χαοτική οικοδόμηση, άναρχη οικοδόμηση, χωρίς το σεβασμό των κανόνων της πολεοδομίας και με πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον αλλά και στις ε, ανθρώπινες σχέσεις. Πρόκειται για μία συνοικία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν η πράσινη συνοικία της πόλης ήταν η πιο πράσινη περιοχή με τα μεγαλύτερα πάρκα, ίσως και η πιο πλούσια συνοικία. τα δημοτικά τέλη είναι εξαιρετικά υψηλά, γι' αυτό και πολλές πολυεθνικές θέλησαν να καταστήσουν την έδρα τους στην γειτονιά αυτή. Πρόκειται όμως για μια γειτονιά η οποία έχει κατά κύριο λόγο διόροφα κτίρια και μία ανάπτυξη την οποία ρυθμίζει με πολύ αυστηρό τρόπο η ε, νομοθεσία. Απαγορεύεται η οικοδόμηση κτίριων που ξεπερνούν τους δύο ορόφους, έτσι ώστε να μην επισκιάσουν τα ιστορικά κτίρια, τα παραδοσιακά κτίρια και μνημεία. Όμως ο Δήμος του πρώτου διαμερίσματος τα τελευταία πέντε χρόνια έχει ερμηνεύσει με έναν τελείως παράδοξο τρόπο την νομοθεσία, δίνοντας τη δυνατότητα σε εταιρείε να οικοδομήσουν μεγαλύτερα κτίρια. Έχει παραβιαστεί λοιπόν εδώ και η κοινοτική νομοθεσία και η τοπική νομοθεσία, αλλά και η ασφάλεια των κτηρίων. Το Βουκουρέστι βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή, επικίνδυνη περιοχή και οι αρμόδιοι μηχανικοί, στατικοί γνωρίζουν ότι τα νέα αυτά κτίρια δεν τηρούν τους κανόνες και την ρουμανική νομοθεσία όσον αφορά την ασφάλεια των κατασκευών. παραδείγματος χάριν όσον αφορά τους ε, χώρους στάθμευσης που πλέον δεν είναι υποχρεωτικά στο υπόγειο αλλά στο ισόγειο ή, ή σε κάποιο όροφο. Αυτό παραβιάζει τους ε, αντισυσμικούς κανόνες και πραγματικά δεν είναι η μόνη παραβίαση. Υπάρχει επίσης και λεύκανση βρώμικου χρήματος, νομοσύπιση, δηλαδή παράνομων εσόδων. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και όσον αφορά τις πληρωμές, τα εμβάσματα, τα τραπεζικά εμβάσματα, καμία απολύτως ρύθμιση δεν έγινε ε, σεβαστή. Όσον αφορά τώρα τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Βλέπουμε ότι το ισόγειο αυτών των κτηρίων έχει πλέον μετατραπεί σε διαμερίσματα και σε και βεβαίως αυτό έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις ε, στο περιβάλλον, επιβαρύνοντας τη μόλυνση της πόλης. Όσον αφορά τώρα τους χώρους στάθμευσης, σύμφωνα με τις άδειε που έχει δώσει ο Δήμος, δεν προβλέπονται σε επαρκή αριθμό. καθότι πολλές φορές βλέπουμε ότι τα υπόγεια έχουν μετατραπεί σε διαμερίσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα αυτοκίνητα δεν έχουν χώρους στάθμευσης. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, καθότι δεν τηρούνται οι κοινοτικές ε, νομοθεσίες, μπορεί να οδηγήσουν και σε ένα επιβαρυντικό πρόστιμο για τη χώρα μου. Τα κτίρια αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον της πόλης. Η μόλυνση σήμερα χαρακτηρίζει τις συνοικίες αυτές και πλήττει ε, τους κατοίκους αυτών των γειτονιών. Σας ζητώ λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να σταλεί και ένα αντίγραφο αυτής της υπόθεσης στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο καθότι η αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών τουλάχιστον για κάποιες από τις πτυχές αυτής της αναφοράς είναι αποδεδειγμένη. Ζητώ επίσης να σταλεί αυτό και στον συνήγορο του πολίτη της χώρας μου γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά και έχει ευαισθητοποιήσει όλους τους κατοίκους του πρώτου διαμερίσματος του Βουκαρεστίου. Σε ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας και είμαι πεπισμένος ότι αυτή η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή και θα την έχουμε υπό επεξεργασία και στη νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει βεβαίως να δούμε ποια είναι η αντίδραση, ποια είναι η απάντηση των ρουμανικών αρχών, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη και σημαντική σειρά παραβιάσεων. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρο. Εγώ το πρώτο που θα έκανα ήταν να απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιγόντως να απαντήσει. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τρούτσα. Δεν είναι μόνο στη Ρουμανία το πρόβλημα, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια έργα που γίνονται σε διάφορες συνοικίες όπου αντιδρά η ίδια η γειτονιά ε, Γι' αυτό μια έκκληση θέλω να απευθύνω στις αρχές. Στην Ισπανία πρόσφατα στην πόλη Μπούργος ε, σε μια συνοικία είχαμε πρόβλημα και τελικά η τοπική αυτοδιοίκηση ε, ανέστηλε την κατασκευή ενός έργου με το οποίο διαφωνούσαν οι πολίτες και υπό την έννοια αυτή και εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Μποστινάρου. Να στείλουμε αντίγραφο και στη Ρουμανική Βουλή αλλά και στο συνήγορο του πολίτη της Ρουμανίας και να αφήσουμε βεβαίως ανοιχτή την αναφορά για να δούμε αν μπορούμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής γρήγορα να δώσουμε απάντηση για να μπορέσει ο κύριος Τρούτσα ο ε, αναφέρον να είναι βέβαιος ότι θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα του. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και να είστε βέβαιος ότι θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Και περνούμε αμέσως στο σημείο 21. Πέντε αναφορές έχουμε σε μία εδώ συγκεντρωμένες. Όλες έχουν να κάνουν με την ενδεχόμενη αδειοδότηση διερεύνηση κοιτασμάτων πετρελαίου στη Φορτεβεντούρα και στο Λασαρότε της Καναρίους νήσους. Είναι πέντε αναφορές που έχουν ομαδοποιηθεί όπως είπαμε. Προτείνω την εξής μέθοδο, να δώσουμε πρώτα το λόγο λογικά ε, στους συντάκτες, ο κύριος Πέντρο Ερνάντεθ Καμάτσο, μετά θα δούμε ένα βίντεο ε, της κυρίας Ελένα Σόλης που απουσιάζει και μετά θα ακούσουμε την κυρία Μαρία Λντεκάρμεν ε, Καμπρέρα Γονσάλης, τον κύριο Ντομίνγκο Μοντανιέθ, συγγνώμη, και τέλος την κυρία Μαρία Μερσέδες Γκόμες Σάντε. Γνωρίζετε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο, έτσι. Σας έχουμε δώσει χρονογόρευσης, μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά οι βουλευτές. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Ε, σας ευχαριστούμε που φέρετε εδώ τη συζήτηση αυτή, η οποία υπερβαίνει βεβαίως κατά πολύ ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα των Καναρίων νήσων. Είναι ένα ζήτημα πανευρωπαϊκό και θα δώσουμε αμέσω το λόγο στον ε, αναφέρον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο και την ευκαιρία να έρθουμε από τα Κανάρια εδώ να σας εξηγήσουμε ένα θέμα που όπως είπατε και εσείς υπερβαίνει ε, το θέμα του νησιού της Πορτεβεντούρα και των ε, Καναρίων είναι πολύ ευαίσθητο και ιδιάζουν το θέμα για τον πλανήτη ολόκληρο. Γίνεται λόγος για την ενέργεια, για το περιβάλλον και το βασικό ζήτημα της ανθρωπότητας που είναι η λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχουν σε αυτή ε, την ε, υπόθεση και γνωρίζουν πόση ευαισθησία υπάρχει. Εμείς ήρθαμε εδώ να ζητήσουμε από την Επιτροπή σας, Επιτροπή Αναφορών, να μάθετε από πρώτο χέρι τι κάνει η Ισπανική κυβέρνηση και πώς μας μεταχειρίστηκαν μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς έδωσαν τις άδειες στην εταιρεία αυτή την πετρελαϊκή να τα γνωρίζετε από πρώτο χέρι, από τη δική μας φωνή για διάφορους λόγους. Πρώτον, διότι έχει ολέθριες ε, συνέπειες ε, και κινδύνους αυτή η υπόθεση. Γνωρίζετε ότι από τις 20 Απριλίου του έτους 2010 υπάρχει ένα πριν και ένα μετά στην εξόριξη πετρελαίου από βαθαία ύδατα. Και ξέρετε ότι αυτό που επέτρεψε η Ισπανική κυβέρνηση για ε, την περίπτωσή μας είναι πάνω από 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχει επιτρέψει σε βαθαία ύδατα ε, πετρελαιοπηγές που είναι αντίστοιχα της έκθεσης όλων των Καναρίων νησιών. Μία πετρελαιοπηγή έχει πάνω από 20% ε, πιθανοτήτων να έχουμε το ίδιο ατύχημα με τον κόλπο του Μεξικού της 24ου ε, του 2010. Δεν τα έχει λάβει υπόψη αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνανε μια ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2010, μετά έγινε σχέδιο κανονισμού τον Οκτώβριο του 2011 και τελικά οδηγία κοινοτική κατέληξε για ε, να ρυθμίζει τις πετρελαϊκές εξορίξεις σε βαθαία ύδατα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στα Κανάρια νησιά αυτό θα γίνει ε, ε, χωρίς να υπάρχει καμία εγγύηση για το παραμικρό. Επίσης, θέλουμε να θέσουμε επιτάπητο στο εξή ζήτημα. Στα Κανάρια νησιά υπάρχει τεράστια κληρονομιά από πλευράς βιοπικιλότητας. Οι ερευνητές, οι επιστήμονες, οι γνώστες του ε, θαλασσίου περιβάλλοντος ε, χαρακτηρίζουν τα Κανάρια το μεγάλο καλάπαγκο του Ατλαντικού και αυτό εμείς θα το θέσουμε σε κίνδυνο. Αυτή η τεράστια βιοπικιλότητα είναι το μοναδικό κεφάλαιο που έχουμε εμείς στις Κανάριες νήσους. Το φυσικό μας περιβάλλον έχουμε με τον τουρισμό μας. 12 ε, εκατομμύρια πολίτες από όλο τον κόσμο έρχονται κάθε χρόνο στα Κανάρια νησιά για τουρισμό ακριβώς λόγω του φυσικού κάλους και τίποτα άλλο. οι μετεωρολογικές δικές μας συνθήκες εκεί και η βιοπικιλότητα είναι ο πλούτος μας. Αυτό λοιπόν το κεφάλαιο κινδυνεύει ε, στο βωμό μιας πολυεθνικής εταιρείας για να κάνει ιδιωτικά κέρδη, ενώ η δραστηριότητα που σήμερα οδήγησε σε βαθιά ε, αλλαγή και μετασχηματισμό τα Κανάρια, ο τουρισμός δίνει φαΐ σε πάνω από 2 εκατομμύρια Καναρίους ε, που ζουν εκεί. Είναι η βασική μας δραστηριότητα ο τουρισμός. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εξόρυξη πετρελαίου στα Κανάρια νησιά εντάσσεται σε ένα ευρύτατο πρόγραμμα που έχει κινήσει η Ισπανική κυβέρνηση. Θα πρέπει να μάθει η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να γνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια η Ισπανική κυβέρνηση πάνω από 1,5 εκατομμύριο εκτάρια στη θάλασσα έχει δώσει άδειες και δεν το ξέρει κανείς. Δεν ακούνε πουθενά τους πολίτες, συγγεί ηχθείω. Ούτε έχουν αξιολογηθεί από πλευράς ε, της κοινοτική οδηγίας που οφείλουν να εφαρμόσουν. 42 του 2001. Τι σημαίνει αυτό. Ότι υπάρχουν και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εφαρμόζουν στην επικράτειά τους και στα πετρελαϊκά τους στη θάλασσα εφαρμόζουν λέγω αυτή την οδηγία. Ε, η Νορβηγία η Μάλτα, η Κύπρος, η Ισλανδία, η Μεγάλη Βρετανία εφαρμόζουν αυτή την κοινοτική οδηγία. Και εμείς εκλυπαρούσαμε επανειλημμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, υποχρεώσει την κυβέρνησή μας να σεβαστεί την οδηγία. Δεν το έπραξαν. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε μια στρατηγική απόφαση τέτοιων χαρακτηριστικών. Γιατί είναι πραγματική απόπειρα Ε, καταστροφής της ζωής μας που το αναγνωρίζει και ε, η νομολογία ε, του δικαστηρίου και η σύμβαση του Άργους το 98 και έχει συνεπογράψει και η Ισπανική κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, σας έθεσα το πλαίσιο και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Ισπανικό κράτος έχει εγκρίνει 1,5 εκατομμύριο εκτάρια λοιπόν για εκμετάλλευση, χωρί συμμετοχή του πληθυσμού, χωρί διαβούλευση και χωρί ελεύθερο ανταγωνισμό. Γιατί όλο αυτό το χρόνο, πάνω από δύο χρόνια, εμείς οικετεύουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να λάβει υπόψη τι καταγγελίε από τι τοπικέ αρχέ, την ισιωτική συνέλευση, την κυβέρνηση των ε, Καναρίων, ε, περιβαλλοντικέ οργανώσει, οργανώσει πολιτών. Γιατί δεν το κάνουν. Γιατί δεν είναι δυνατόν, γιατί είναι ειδική περίπτωση τα Κανάρια ας πούμε, να υπάρχει τέτοια δραστηριότητα χωρίς να έχουμε δει άλλες εναλλακτικέ. Έχουν ξεχάσει το κεφάλαιο ένα, το άρθρο μάλλον ένα αυτής της οδηγίας θα πρέπει πάντα να μελετώνται οι διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις σε κάθε σχέδιο, σε κάθε οικονομικό και ενεργειακό μοντέλο που θέλει κανείς να εφαρμόσει σε μια περιοχή. Θα πρέπει να γνωρίζει η Ευρώπη ότι τα Κανάρια νησιά μπορεί να είναι το παγκόσμιο παράδειγμα για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε και έδαφος, έχουμε συγγνώμη, και ήλιο ε, και ε, αέρα και ε, παλήρια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανανέωση και όχι την εξόριξη των ορυκτών καυσίμων. Η πολυεθνική αυτή μιλάει για 20 χρόνια για την ε, εκμετάλλευση. 20 χρόνια δραστηριότητες άμα αρχίσουν ε, να εξορίσουν εκεί πετρέλαιο. Η γεωργία, η αλληλεία, ο τουρισμός, η φυσική πόρη ε, στα Κανάρια μπορεί να είναι ε, ένα μοντέλο αηφόρου ανάπτυξης και αέναης ανάπτυξης, αν ξέρουμε να το κάνουμε σωστά, γιατί να το διακινδυνεύσουμε αυτό το μοντέλο, τον τρόπο ζωής, απέναντι σε μια δραστηριότητα που ξέρουμε ότι είναι εξορυκτική, ότι είναι πεπερασμένη χρονικά ε, και έχει και κίνδυνο σε πολύ βαθιά ύδατα και ε, η πετρελαϊκή βιομηχανία δεν έχει λύσει τίποτα σε αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει η Επιτροπή σας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ξέρει όλα αυτά. Μας έχει απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις κοινοβουλευτικές και έχει πει τα εξής. Πρώτον, η οδηγία του 85 που τώρα είναι 2001 παραγνωρίζει το παράρτημα 2, 3, 1 κτλ ε, λέει ότι εξαιρούνται από αυτή την οδηγία. Καθόλου δεν εξαιρούνται. Και ε, δεν κάνει καμιά διάκριση ανάμεσα στη διερεύνηση για πετρέλαιο και στην εξόριξη. Από την άλλη λένε, ε, ο κύριος Ποτώνη στις διάφορες ερωτήσεις που κάναμε, από τη μια λέει ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και μετά έρχεται να το ανατρέψει αυτό και λέει ότι έχουν γίνει. Ναι λοιπόν λέει. Και μετά ξαναείπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η άδεια που έχει δοθεί το τελευταίο βασιλικό διάταγμα 16 Μαρτίου 2012 δεν θέτει πλαίσιο για μελλοντική εξόριξη. Ε, είναι διερεύνηση ακόμα. Αυτό που δεν ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το περιεχόμενο του βασιλικού διατάγματος, το οποίο βασίζεται σε ένα έγγραφο που της έφερε η εταιρεία Repsol στις 7 Μαΐου του 2004, που ήδη μιλούν όχι για διερεύνηση, αλλά για ένα σχέδιο πολύ καλά κατηρτισμένο. Εμείς πραγματικά οικετεύουμε, εκλυπαρούμε την Επιτροπή σας να διερευνήσετε για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τελευταίο 1,5 χρόνο μας απαντάει στις ερωτήσεις ε, με τρόπο πώς να το πω, υπεκφεύγει. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και πολύ επικίνδυνα. Και ένα τελευταίο για να μην σας κουράσω. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στα θεμελιώδη δικαιώματα και θέλουμε να το θέσουμε υπόψη σας και αυτό. Η έγκριση για τις διερευνητικές... Ε, α, εδώ είναι κάτι σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει και αντισυσμική προστασία. Είναι σεισμογενής η περιοχή και υπάρχει βιοπικιλότητα τεράστια. Έχουμε πάνω από 30 είδη ε, κοιτών ε, που ζουν εκεί σε αυτά τα ύδατα. Πάνω από 30 Λοιπόν, είναι σεισμογενής το ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού ήταν σε διερευνητικό στάδιο, δεν ήταν εξόριξη. Ε, τους ε- έφυγε ε, ε, εκεί το ε, με διαρροή από την ε, πετρελαιοπηγή στο στάδιο της διερεύνησης, όχι της εξόριξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αξιολογούμε μόνο την επόμενη φάση, όχι τη διερεύνηση, αλλά την ουσιαστική εξόριξη. Ε, λοιπόν, για τα θεμελιώδη δικαιώματα έλεγα, υπάρχει ένα ζήτημα ότι μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να περάσει χωρίς να ρωτηθεί ο πληθυσμός ο οποίος στήγεται άμεσα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά σημαντικό κάτι τέτοιο για να ε, αφαιθεί ε, στα πλαίσια του εμπορίου, δεν είναι μια μπίζνα μεταξύ ε, της πετρελαϊκής εταιρείας και της ισπανικής κυβέρνησης. Έχουμε βουλή, κυβέρνηση τοπική, νησιωτικές συνελεύσεις, επιστημονική κοινότητα και πολίτες που επανειλημμένα εκφράζουν την άρνησή τους. Και αυτή την παραγνωρίζει η κυβέρνηση. Αν μου επιτρέπετε η συνάδελφός μου Έλενα Γιάννης ε, δυστυχώς απουσιάζει αλλά έχουμε ένα βίντεο που θα θέλαμε να δείτε γιατί είναι πραγματικά επιστήμονες που ε, γνωμοδοτούν ή εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για το χρόνο που σας έφαγα. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν να δούμε το βίντεο. Έχετε το κείμενο γιατί δυστυχώς δεν θα μπορέσει ε, να υπάρξει ταυτόχρονη διερμηνία στην ταινία και όσοι δεν μιλάτε ισπανικά Έχετε σε διάφορες γλώσσες τη μετάφραση του κειμένου. Richard Steiner. I'm in Anchorage, Alaska. I was a marine science professor at the University of Alaska for 30 years, specializing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 Βλέπετε λοιπόν ότι τελειώσαμε το βίντεο. Ε, έχουμε τον κύριο Βίλκενς ακόμα από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, τελευταίο, που έχει μελετήσει στο Λανσαρότε 30 χρόνια την ε, χλωρίδα και την πανίδα. Μπορείτε να το βρείτε γραπτό στο κείμενο. Έχουμε χρόνο τώρα, δεν μπορούμε να δούμε το βίντεο. Αναγκαστήκαμε να ε, κόψουμε την ταινία για να ακούσουμε τους παρόντες ε, υπολείπους που δεν έχουμε ακούσει. Θα δώσουμε λοιπόν αμέσως το λόγο στους παρόντες, αλλά παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Έχουμε πάρα πολύ αυστηρό θέμα με το χρόνο. Ε, η κυρία Μαρία Ντελκάρμεν Κάμπερα Μεσάλες και ο κύριος Μοντάνιεθ θα πάρει το λόγο να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα ε, για αξιοπρεπή ζωή για όλα τα παιδιά του κόσμου που ζουν στο Λασαρότη και τη Φορτεβεντούρα. Για τους γονείς και παππούδες μας που αγωνίστηκαν να ζούμε αξιοπρεπώς σε αυτά τα νησιά και για τις επερχόμενες γενναίες. Γι' αυτό εγώ καταγγέλω και σας παραπέμπω στην αναφορά μου. Αυτό το δικαίωμα κυρίες και κύριοι είναι υποσοβαρή απειλή από την κυβέρνηση της Ισπανίας που ε, στα ύδατά μας ε, το νερό που πίνουμε έχουν επιτρέψει τις ε, Θα πρέπει να ε, ξέρετε και να μην ξεχνάτε ότι ο μοναδική πηγή για μας πόσιμο νερού είναι η θάλασσα. Δεν έχουμε ούτε ποτάμια ούτε λίμνες και η βροχή ε, πέφτει λίγη. Και θα πρέπει να καταλάβετε ότι η απόφαση που θα πάρει η Ευρώπη θα είναι η εικόνα που δίνει η Ευρώπη στον κόσμο. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά θεωρώ ασύλληπτο στον 21ο αιώνα ένα ευρωπαϊκό έδαφος όσο μακριά και είμαστε από την Ήπειρο να είμαστε χωρίς πόσιμο νερό όταν η Ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε το βασιλικό διάταγμα 547 του 2012 παραβίασε από τη συνθήκη της Ένωσης το άρθρο 74 που ορίζει ως βασική αρχή τη διατήρηση, αφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλά στο πρώτο της άρθρο για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που είναι απαραβίαστη συν την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα στο πνεύμα όπως και στο γράμμα και στο στόχο της. Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα κυρίες και κύριοι ε, να σας αναφέρω την πρώτη παράγραφο που λέει ότι το νερό δεν είναι ένα εμπορικό αγαθό αλλά είναι κληρονομιά που θα πρέπει να ε, προστατεύουμε. Δίνουν τώρα το νερό όλου του κόσμου και των τουριστών σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Για να σας δώσω ένα στοιχείο που κατά την άποψή μου θα πρέπει να σταματήσει το πρόγραμμα αυτό. Στο άρθρο 14 ορίζεται υποχρέωση διετίας ε, ε, έκθεση ε, στο κοινό σε διαβούλευση για οτιδήποτε σημαντικό γίνει σε σχέση με το νερό που πίνει ο κόσμος από την αφαλάτωση. Και ξέρετε πόσο μας έδωσε η κυβέρνηση. Ένα μήνα και 20 μέρες αν θυμάμαι καλά και μάλιστα αυγουστιάτουκα για ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου το νερό που για μένα είναι πολύ σημαντικό Οχτώ σελίδες αναφέρουν, οχτώ σελίδες με καμία λύση να προτείνεται για το τι θα συμβεί στα νησιά μας εάν γίνει ε, καμία διαρροή στο νερό. Η Ισπανική κυβέρνηση απαντάει λοιπόν και μας λέει, όπως ακούσαμε προηγουμένως, ότι σε περίπτωση διαρροής ε, θα αναλάβουν οι τοπικές αρχές την υδροδότηση του πληθυσμού. Μα οι τοπικές αρχές έχει μαλλιάσει γλώσσα τους να απορρίπτουν αυτό το σχέδιο παραγνωρίζουν και αγνοούν και τον εσωτερικό μας κανονισμό λειτουργίας και το κοινωτικό. Ο Υπουργός Βιομηχανίας διαβεβαιώνει ότι θα αρχίσουν το Μάιο εξορίξεις ε, χωρίς να έχουν απαντήσει σε χιλιάδες ενστάσεις ε, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δεν δίνει λύσεις για το νερό. Παραγνωρίζει και αγνοεί και την Ισπανική νομοθεσία και την κοινωτική νομοθεσία. αυτό το δίλημα πόσιμο νερό ή πετρέλαιο από ό,τι φαίνεται είναι άλυτο, μα δεν είναι καν δίλημα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονα, ούτε τεχνικέ γνώσει έχω, αλλά είμαι πολίτη και μπορώ να σα πω και η ιστορία με δικαιώνει και έχω δικαίωμα να ερωτώ. Δείχνει λοιπόν η ιστορία ότι ακόμα και μια ελάχιστη διαρροή οι μονάδε αφαλάτωση παραλύουν και μας μένουν οι πολίτε, ε, τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσει η κτηνοτροφία, η γεωργία χωρί νερό καθόλου. Δεν έχουμε σύστημα αποθήκευση υδάτων. Ακόμα και αν γίνει κανένα θαύμα και δεν υπάρχει ε, διαρροή, αφήστε που δεν πιστεύω στα θαύματα, πόσο μάλλον εδώ, ε, θα ε, έχουμε καρκινογόνο μόλυνση στο νερό μας. Παράδειγμα, πώς δρούν ορισμένε εταιρείε στη Νότια Αμερική. Το έχουμε δει σε εκθέσεις της Greenpeace και άλλων που σας έχουμε θέσει υπόψη εδώ στο Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, επιτρέπετε αν ε, να γίνει μια τέτοια εξόριξη. Θα το κάνατε σε ένα ταμιαυτή νερού, ε, σε μια τεχνητή λίμνη υδροδότησης μιας μεγάλης πόλης ε, στην υπηρετική Ευρώπη. Σκεφτείτε μας και εμάς, ακόμα και αν είμαστε πιο κοντά στην Αφρική από ότι στην Ευρώπη. Μέχρι και σε 10 χιλιόμετρα από τη μονάδα αφαλάτωσης είναι η πιο κοντινή πετρελοπηγή είναι στα 9,5 χιλιόμετρα, ακόμα και αν λένε ότι είναι στα 60 η Ρεψόλ. Και ε, παρακαλώ να το σκεφτείτε αυτό. Κοιτάξτε, Στη δεκαετία του 70 έγινε μεγάλη αλλαγή στα νησιά μας Λανσαρότε και Φορτεβεντούρα. Κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, δημογραφική ανάπτυξη. Φτάσαμε πιο κοντά στον κόσμο. Το γεγονός ότι είμαστε σήμερα εδώ το οφείλουμε στη μονάδα αφαλάτωσης που μας επέτρεψαν ε, οι γονείς μας ε, χάρη στην πρόοδο να πάμε να σπουδάσουμε και να έρθουμε μέχρι εδώ. Ε, σήμερα είναι τελείως ηλικιώτης η κατάσταση. Μας έχουν εγκαταλείψει οι κεντρικές αρχές της Ισπανίας παρόλο που όλες οι τοπικές αρχές, η κυβέρνηση των Καναρίων και ο πληθυσμός έχει αντιταχθεί 100%. Γι' αυτό σας λέγω ότι είμαι πεπισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο θεσμός σας εκπροσωπεί την καλύτερη εγγύηση για το δημοκρατικό μας σήμερα σύστημα, γι' αυτό ήρθα κιόλας. Σας παρακαλώ σταματήστε αυτό το τρελό πρόγραμμα και σκεφτείτε τη Σύμβαση των, Ηνωμένων ε, Εθνών για την προστασία των υδάτων, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 12 και στην αιτιολογική σκέψη 35 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ήδατα, που ορίζει ότι είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένας συντονισμός και με το Μαρόκο για να προστατεύουμε τα νερά μας. Γιατί ε, και στα χωρικά ύδατα του Μαρόκου μπαίνουν. Ευχαριστώ πολύ και θα δώσω το λόγο στο χημικό μηχανικό συνάδελφο που θα σας εξηγήσει τα τεχνικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δον Ντομίνκο, Μοντάνιες Μοντάνιες. Παρακαλώ να τηρήσετε, αν γίνεται, το χρόνο σας. Καλημέρα σας. Θα προσπαθήσω στο δίλεπτο που μου δώσατε να σας πω πώς έχει η κατάσταση στη Φορτοβεντούρα από την τεχνική σκοπιά και προσωπικά προσπαθώ να σας διαβεβάσω τον πιθανό κίνδυνο που υπάρχει σε περίπτωση που υπάρξει πετρελοκυλίδα μεγάλης κλίμακας. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί μια χημική αντίδραση τέτοιας διάστασης ε, να λάβει χώρα χωρίς να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Η Φορτεβαντούρα από γεωγραφικής απόψεως δεν έχει φυσικούς πόρους έτσι κι αλλιώς επιφανειακή ύδατα δεν έχει, είναι σχεδόν έρημος, δεν, δεν βρέχει. Και τα υπόγεια ύδατα είναι χειρίς της ποιότητος. Αφήστε δε που είναι και πάρα πολύ λίγα. Δεν μπορούμε καμιά στιγμή να σκεφτούμε ότι μπορούμε να αντλήσουμε ύδατα από το υπέδαφος. Έχουμε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τη μάζα του νερού, του υπογείου ύδατος, ε, σε καλή κατάσταση και ποσοτική και χημική. Τι σημαίνει αυτό μοναδικός μας πόρος ε, για υδροδότηση είναι η θάλασσα. Η βιομηχανική παραγωγή, αφαλάτωση, από εκεί παίρνουμε το πόσιμο νερό. Το 100% είναι από τη θάλασσα, από βιομηχανική παραγωγή. Αν δεν είχαμε εμείς τις μονάδες αφαλάτωσης, δεν θα είχαμε πόσιμο νερό. Ξέρουμε ότι είναι μια τεχνολογία ε, ε, πολύ ε, διαδεδομένη στον κόσμο, έχει μεγάλη απόδοση και καλή και τα Κανάρια νησιά είναι και αναφορά για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτές οι εγκαταστάσεις είναι διασπαρμένες στην ανατολική ακτή της Φουερτεβεντούρας και αντλούν τα ύδατά τους από μικρό έδαφος, μικρό βάθος, συγγνώμη. τι θέλω εγώ να σας πω αν αρχίσει τώρα και εξοεκτική δραστηριότητα του μεγέθους και της κλίμακας που φιλοδοξούν, θα πρέπει να είναι εγγυημένη η κάλυψη της ζήτησης σε νερό. Γιατί σε περίπτωση διαρροής και πετρελοκυλίδας ε, θα χαλάσουν οι ε, εγκαταστάσεις, τα εργοστάσια αφαλάτωσης ανάλογα με την πετρελοκυλίδα και μπορεί μέχρι και οι να σταματήσουν. Δηλαδή δεν θα έχουμε νερό είναι περιορισμένη η υδραυλική ε, υποδομή, η αυτονομία, ε, οι σωλήνες υδροδότησης και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τι εννοώ δηλαδή. Μια τέτοια εξορυκτική δραστηριότητα δεν δίνει τα ε, απαραίτητα εχέγγυα σε αυτό το ζήτημα ε, σε σχέση με τα έγγραφα που έχω δει. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το Λασαρότε και για τη Φουέρτεβεντούρα. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί σε περίπτωση διαρροή που δεν ξέρουμε τι μέγεθος θα έχει και τι έκταση, ε, δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς νερό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίος τελευταία μάλλον, η Δόνια Μαρία Μερσέδης Γκόμες Άντεκ. Παρακαλώ και εσείς να τηρήσετε τα δύο λεπτά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ερχόμαι ως ανεξάρτητη πολίτης εδώ, αλλά και μία από τις πρώτες που έχω σπουδάσει θέματα περιβάλλοντος, δεν θα μπω σε θέματα που ανέφεραν οι προλαλήσαντες, θα είμαι σύντομη. Αυτό που ήθελα εγώ να τονίσω και από την προηγούμενη αναφορά είναι η συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση. Και στο γενικό σχεδιασμό. Με την κατάσταση που έχει προκύψει, Θέλω να σας ρωτήσω τι τις έχουμε όλες αυτές τις συνθήκες, ευρωπαϊκές συμβάσεις, προγράμματα τοπικού σχεδιασμού, προγραμματισμού, αν πολλές φορές παίρνονται αποφάσεις σε κρατικό επίπεδο, παραγωνίζοντας τελείως όλες τις δημοκρατικές αρχές που αναφέρουν τα ωραία μας έγγραφα. Συγκεκριμένα, το τοπίο στη Λανσαρότα και το Φορτεβεντούρα είναι εξαιρετικής ευαισθησίας όσο και ιδιαιτερότητας Ε, είναι στο κέντρο άνθρωπος και η φύση. Έχουμε και ε, ε, προστατευόμενες περιοχές της βιόσφαιρας, της UNESCO. Βασίζεται η ανάπτυξή μας κυρίως στον τουρισμό και μάλιστα τον αηφόρο και το βιώσιμο. Και θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα που είναι σε πλήρη ασυμβατότητα με την εξόρυξη πετρελαίου. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο, για τη χωροταξία ε, και νομίζουμε ότι είναι ένα καλό εργαλείο για να προστατεύσουμε το τοπίο μας. Και είναι ποιότητα ζωής, ευημερία και τέτοια θέματα που διακυβεύονται. Δεν υπήρξε καμία διαβούλευση κατά τη λήψη των αποφάσεων, συνεργασία με τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντική απόφαση για το μέλλον μας και δεν μας ερώτησαν. Και εδώ ήρθαμε να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Συνεργασία να επέμβεται σε αυτό το θέμα, παρακαλώ. Και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη νομοθεσία στα Κανάρια νησιά, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός, η Γενική Χωροταξία αποφασίζεται ε, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τον τουρισμό. Στην αιτιολογική έκθεση καταλαβαίνουμε ε, ότι ε, αντιτίθεται το συγκεκριμένο έργο με τις δικές μας κατευθυντήριες γραμμές που είναι η βιώσιμη και η φόρος ανάπτυξη για τα νησιά που να σέβεται το περιβάλλον, το τοπίο, την φυσική κληρονομιά και γενικότερα την επικράτειά μας. Οι αρχές επέμβαση λέγουν ότι επεμβάσεις και οι παρεμβάσεις ιδιωτικές και δημόσιες στο αρχιπέλαγος των Καναρίων θα πρέπει να σέβονται και να διαφυλάσσουν τη φύση, το περιβάλλον, τους πόρους κτλ. κτλ έτσι ώστε οι σημερινές και αυριανές γενιές να μπορούν να υποφελούνται από την κατάσταση αυτή. Ε, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του περιβάλλοντος, πλήττεται σφόδρα. Υπάρχει αρχή της προφύλαξης, η αρχή της αφιβολίας σε αυτά τα θέματα και ε, είναι πολύ οι άγνωστοι και οι άγνωστες ε, πτυχές ε, ως προς τις βλάβες που μπορεί να προκληθούν και μάλιστα ανεπανόρθωτες ζημίες. Ε, και είναι ένα θέμα μεταξύ διαφόρων γενναίων. Δεν θα πρέπει να καταστρέψουμε το περιβάλλον μας ε, για τις επόμενες γενιές. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χρήσης και ωφέλους ε, με δίκαιο τρόπο για όλους τους κλάδους της κοινωνίας και να έχουμε υπόψη μας και τις ανάγκες των μελλοντικών γενιών este es el decreto del 27-2004 Το 2004 έχουμε το διάταγμα 27 ε, για τη χωροταξία του τοπίου και του περιβάλλοντος. Κανονικά ε, υπάρχει μια διετία για την έγκρισή τους από το 2003 και μετά και μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, αλλά έκτοτε δεν έχουμε καμία είδηση. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από το νησί μας και τέλος θέλω να σας ζητήσω εκτός από τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, να φροντίσετε να τηρούνται οι νόμοι για το περιβάλλον και το τοπίο και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, Πρόεδρος. Πριν αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση, θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αγγέλ Φερνάντες Κόμες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε γνώση αυτού του θέματος ε, μέσω πολλών καταγγελιών και διαφόρων αναφορών που έχετε λάβει κι εσείς και μας έχετε διαβιβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια άρχισε μια διερεύνηση του θέματος που όπως είναι λογικό περιορίζεται στις αρμοδιότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή να βεβαιωθούμε ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έχουν σεβαστεί ε, τις διάφορες αρχές και υποχρεώσεις που ισχύουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκουν εφαρμογή σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να πούμε εδώ πρώτα απ' όλα ότι η αρμοδιότητα για την εκμετάλλευση και για την αδειοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων διερευνητικών για τους φυσικούς πόρους εναπόκειται αποκλειστικά ε, στις αρχές των κρατών μελών. Βέβαια, ασκώντας αυτές τι αρμοδιότητές του, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σέβονται ανά πάσα στιγμή τι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που βρίσκουν εφαρμογή ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Έτσι, θα περιορίσουμε ε, τους ενδεχομένους κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες. Τα γνωρίζει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διερεύνησης που σας ανέφερα προηγουμένως, ήρθε σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε τις παρατηρήσεις τους για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σχετικά. Και επίσης ζητήσαμε λεπτομέρειες για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν ε, με σκοπό την τήρηση αυτών των νομοθετικών διατάξεων, την προστασία της φύσης του περιβάλλοντος και ε, τα λοιπά ζητήματα που τυχόν αφηγούν από αυτή την εκμετάλλευση. Οι Ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα σχέδια διερεύνησης ύπαρξη υδρογονανθράκων γύρω από τα Κανάρια νησιά εντάσσονται σε μια μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου και με βάση αυτή ε, επιτραπεί η διερεύνηση, η περιγραφή και η ανάλυση των αμέσων όσο και των εμέσων συνεπειών στο περιβάλλον των διαφόρων δράσεων. Αυτή η ε, διαδικασία είχε και δημόσια διαβούλευση. Είχαν την ευκαιρία όλοι οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν ε, τις απόψεις τους για να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες αρχές. Πριν δοθεί η τελική έγκριση στο έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υπόψη της τίποτα σχετικό με την έγκριση. Δηλαδή δεν έχουν εγκριθεί ακόμα τα προγράμματα στα οποία αναφέρονται οι αναφορές αυτές. Δεν έχει ε, εκδοθεί η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αποφανθεί λοιπόν ε, αν ε, όχι, έχει υπάρξει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου μέχρι να δοθούν οι εγκρίσεις και οι ε, μελέτες. Όσο είναι ακόμα καθοδόν αυτή η διαδικασία, το μόνο που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να απαιτεί σχολαστική τήρηση των κανόνων που ισχύουν. Από τη στιγμή που θα δοθεί η έγκριση θα ε, παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δραστηριότητες ε, της Ισπανικής κυβέρνησης έτσι ε, ώστε να βεβαιώνεται ότι τηρείται ισχύουσα νομοθεσία. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ομιλητές τώρα, συναδέλφους που θα πάρουν το λόγο, τους εξή τέσσερις, πέντε, καλά, εντάξει. Με τη σειρά όλοι θα μιλήσετε. Εγώ θα μιλήσω με διπλή ιδιότητα. Μία την προσωπική μου και δεύτερη του Προέδρου για να κάνω ε, τις ε, τελικές παρατηρήσεις. Ο κύριος Λόπες Αγγιλά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ είναι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, και πρωταγωνιστούν οι αναφέροντες εκπρόσωποι των πολιτών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ιστού που έρχονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαλούμενοι κοινοτικό δίκαιο και ζητώντας από τα θεσμικά όργανα να φροντίσουν να διατηρηθεί. Ε, είναι δουλειά λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της Εκτελεστικής. Άκουσα τους αναφερόμενους και θέλω να πω ότι υποστηρίζω και η ομάδα μου και η Ισπανική Αντιπροσωπεία, η Σοσιαλιστική ε, ομάδα, η σοσιαλιστική αντιπροσωπεία, ε, ανεπιφύλακτα συμμερίζομαι ε, τις αμφιβολίες και τις αγωνίες των όσων ακούσαμε. Θα επικεντρωθώ εγώ λοιπόν στο εξής. για το κατά πόσο τηρείται η κοινωνική νομοθεσία. Στο Βασιλικό Διάταγμα 47 το 2012 κανονικά θα πρέπει να γίνει συζήτηση, διαβούλευση για τις αντιθέσεις. Έχουμε μια στρατηγική για τις ανανεώσιμες, καθαρές και βιώσιμες και αηφόρες μορφές ενέργειας. Αυτό θα πρέπει να προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια η Ισπανική κυβέρνηση. Επίσης πρέπει να πω ότι έρχεται αυτό σε αντίφαση με το μοντέλο αηφόρου βιώσιμου τουρισμού που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνίας στα Κανάρια νησιά. Επίσης, δεν θα αναφερθώ στην περιφρόνηση προς τους πολίτες. Επανειλημμένα έχουν εκφράσει και τα θεσμικά όργανα, ε, η κυβέρνηση των Καναριών, η Βουλή των Καναριών και οι νησιωτικές συνελεύσεις των δύο νησιών που θίγονται περισσότερο από αυτή την έγκριση που είναι η Λανσαρότη και η Φορτεβερτούρα. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά στην άκρη. Δεν θα αναφερθώ σε όλα αυτά ε, που αφορούν την πολιτική στα Κανάρια νησιά και στην Ισπανία γενικότερα. Θέλω όμως να επικεντρωθώ σε αμφιβολίες ως προς την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας. Η κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η προστασία, η οδηγία 2011 κάθετος 92 για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος. 92-43, άλλη οδηγία που αφορά τη διαφύλαξη των οικοτόπων ε, των ε, αγρίων ειδών ε, χλωρίδας και πανίδας και των δασικών ειδών. Έχουμε καμιά δεκαριά εκεί φυσικά πάρκα και προστατευόμενες περιοχές που είναι και τμήματα ε, της Natura 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από την ε, ε, θαλάσσια ζώνη των Καναρίων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και την έχει χαρακτηρίσει έτσι ο IMO. Ένα άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται πολύ συχνά έχει να κάνει με την έλλειψη ανταγωνισμού. Δηλαδή, σε αυτή την παραχώρηση προς αυτή την εταιρεία είναι μία η εταιρεία. Δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Άρα αμφισβητείται και η οδηγία 94 κάθετος 22 που έχει να κάνει με τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ και μπορεί να είναι ανεπαντόρθωτος οι συνέπειες. Είχαμε δει όταν αρνήθηκαν να δώσουν την πρώτη άδεια το 2001 γιατί υπήρχε δυνατότητα ε, πετρελοκυλίδας. Το είδαμε να συμβαίνει αυτό στο 2011 ε, στον κόλπο του Μεξικού με ε, μία ακτίνα ε, ζημιών 250 χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το Λανσαρότε και την Φορτεβεντούρα που είναι πιο κοντά από 60 χιλιόμετρα σε αυτό το πολύτιμο περιβάλλον που πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε. Ο κίνδυνος είναι δεδομένος και δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι η τελική άδεια θα ε, τηρεί σχολαστικά την κοινοτική νομοθεσία. Γι' αυτό οι σοσιαλιστές ζητούν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά για να βεβαιωθούμε ότι όλες αυτές ε, οι ε, καταγγελίες, οι ισχυρισμοί, τα παράπονα κτλ. να ληφθούν υπόψη. Πάει η Ισπανική κυβέρνηση και δίνει το έργο σε μία και μοναδική επιχείρηση. Αυτή την εγγύηση δεν την έχουμε σήμερα. Ξέρουμε ότι δεν τηρήθηκαν οι ε, προθεσμίες. Καλοκαιριάτικα βάλαν μια προθεσμία εκεί έτσι ώστε μέσα στη θερινή ραστόνη να το περάσουν άρον άρον. Και σας μεταφέρω εδώ τη σημασία του θέματος. Η σοσιαλιστική ομάδα, επαναλαμβάνω, ζητεί να παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Και αναφορά. Ευχαριστώ. Ξέρετε, έξι έχετε ζητήσει το λόγο συνολικά. Θεωρητικά δωδεκάμιση το σφυράμε. Γιατί θα μείνουμε από διερμηνία. Παρακαλώ να αυτορυθμιστείτε κάπως για να μιλήσετε όλοι εντός των πλαισίων της διερμηνίας. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Μποστινάρο που είχε ζητήσει πρώτο το λόγο και το είχαμε ξεχάσει. Παρακαλώ έχετε το λόγο και μετά οι υπόλοιποι. Thank you very much. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και δεκαετίες οι πετρελαϊκές εταιρείες συνεχίζουν να ζητούν την εκμετάλλευση. Αυτό που τουλάχιστον σήμερα ξέρουμε, είναι ότι συνέβη αυτό που συνέβη, αυτή η τραγωδία στον κόλπο του Μεξικού. Γνωρίζουμε σήμερα τις επιπτώσεις. Η BP, μια γιγαντιαία βρετανική επιχείρηση, δημιούργησε αυτή την καταστροφή στην Αμερική. Καταλαβαίνετε ότι το μέγεθος αυτής της καταστροφής είναι αδύνατον να περιοριστεί σήμερα. Και ελπίζω, ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία και να μάθει από αυτό το πάθημα. Εδώ όμως δεν βλέπω τίποτα όσον αφορά τα συσσωρευτικά αποτελέσματα, τα συσσωρευμένα συγγνώμη αποτελέσματα. Δεν βλέπω πουθενά να γίνεται αναφορά για μία αξιολόγηση των επιπτώσεων για το περιβάλλον. Πρόκειται για πολύ βαθιά νερά με μεγάλη βιοπικιλότητα προστατευόμενη από το πρόγραμμα Natura 2000. Πρόκειται επίσης για μία περιοχή που εξαρτάται από μία μόνο πηγή πόσιμου ύδατος που είναι η θάλασσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία αξιολόγηση είτε στρατηγικός σχεδιασμός. Και την ίδια ώρα αναρωτιέμαι που είναι ο τριμερής διάλογος μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πού είναι η διαφάνεια, πού είναι η αντικειμενικότητα, πού είναι η ουδέτερη στάση έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο σχέδιο. Όταν ξεκίνησε αυτό το σχέδιο από την επιχείρηση Repsol, υποβλήθηκε μία μελέτη η οποία αυτονομάστηκε ουδέτερη και αντικειμενική. Μα αυτό είναι αστείο, αστείο. Ποια είναι η συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών, πού είναι οι τοπικές αρχές, πού είναι οι τοπικοί βουλευτές, Όλοι ήταν αντίθετοι με αυτό το σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ μας λέει ότι υπήρξε πραγματική διαβούλευση όλων των εμπλεκόμενων μερών. Μα αυτό είναι δεύτερο αστείο, θλιβερό αστείο θα έλεγα. Και ανεπαρκής απάντηση από μέρους της Επιτροπής. Τέλος, πού είναι οι εναλλακτικέ λύσεις, οι οποίες είναι προαπαιτούμενο όσον αφορά την ε, τροποποίηση της ε, οδηγίας. Δεν υπάρχουν εναλλακτικέ προτάσεις ούτε όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Πραγματικά λοιπόν θα συμφωνήσω εδώ πλήρω με τον Χωσέ Λόπες Αγγιλάρ. Η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή υπό την ε, παρακολούθηση, την αυστηρή παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμείς η Επιτροπή Αναφορών είτε οι διάδοχοί μας θα πρέπει να εξετάσουν με μεγάλη προσοχή όλα όσα συμβαίνουν στις Κανάριες νήσους. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, η Ισπανία θέλει να καταστρέψει ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των νησιών αυτών ή θέλετε πραγματικά να αυτή η περιοχή, να πληγεί από μια καταστροφή που απορρέει από την πετρελαϊκή εκμετάλλευση. Κύριο Μάτο, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Υποστηρίζω απολύτως και σέβομαι εκείνους που ήρθαν και μίλησαν εδώ πως θα γινόταν διαφορετικά άλλωστε. Βέβαια, ο σεβασμός αυτός δεν σημαίνει υποστήριξη των ισχυρισμών τους και των φιλοδοξιών. Ε, ακούσαμε πολλά πράγματα. Σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να ακούσει κανείς πολλά άλλα. Μπορεί να κάνει πολιτική, μπορεί να δημαγωγεί, μπορεί να λαϊκίζει, μπορεί να μιλάει και για νομιμότητα. Βασικά αυτό πρέπει να κάνει η δική μας ε, επιτροπή. Έκαναν αναφορές οι άνθρωποι, ήρθαν να μας ενημερώσουν, να καταγγείλουν για μια σειρά ε, παραβιάσεων ορισμένων οδηγιών. Εγώ κρατώ αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει όλο μου το σεβασμό παρά τα όσα είπε ο προλαλή σα, είπε ότι δεν έχει παραβιαστεί μέχρι στιγμή καμία νομοθεσία. Έτσι έχει η πραγματικότητα. Θα είχα κι εγώ πολλά επιχειρήματα για να αντικρούσω αυτά που ακούσαμε ή να προσπαθήσω τουλάχιστον ε, ε, για τις ε, παραβιάσεις και ορισμένων οδηγιών. Δεν θα το κάνω, κυρίως γιατί δεν έχω χρόνο και επίσης γιατί δεν έγινε καμιά ανάλυση σε βάθος για αυτές τις εικαζόμενες ε, παραβιάσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν υφίστανται. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δώσω μια στοιχειώδη ιδέα. Περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για φέτος και για πέρσι και δεν κοιτάμε ιστορικά τι έχει γίνει και τι λέει η ιστορία. Ότι αυτή η παραχώρηση και η άδεια είναι συνέχιση προηγούμενης αδείας του έτους 2001. Παράταση είναι, δεν είναι νέα έγκριση αδείας. Απλώς ε, συνέχιση της αρχικής παραχώρησης που λύγει. Και δεν υπήρχε, όπως είπαν τα δικαστήρια τότε, ε, την ε, σωστή περιβαλλοντική προστασία. Ωραία. Ε, από πέρσι άρχισε αυτή η συζήτηση θα γίνει δημόσια διαβούλευση. Η περιβαλλοντική μελέτη θα μπορούσε να είχε γίνει με τρόπο πολύ λιγότερο αυστηρό. Δεν είχε τις απαιτήσει αυτές που ε, ακολούθησε η εταιρεία. Ήταν πιο αυστηρός ο έλεγχος, δημόσια διαβούλευση για να συμμετέχουν. Βεβαίως και πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες. 5.169 αιτήματα ε, ε, έχουν διαβιβαστεί όλα στο σύνολό τους αρμοδίως και εμείς μπορούμε να πούμε ότι έχουν ληφθεί όλα υπόψη. Αυτή η δημόσια διαβούλευση επιπλέον έφτασε σε όλα τα θεσμικά όργανα, ε, σε πανεπιστήμια, Ινστιτούτο Οκεανογραφικό, ε, Ενώσεις ε, Αλλιέων, ΜΚΟ, Λιμάνια, γενικές συνελεύσεις νησιωτικές μέχρι και κάτι ε, οργανώσεις για την πράσινη ποδηλασία για να καταλάβετε. Ε, σε όλους έφτασε τους αποδέκτες ε, αυτή η διαβούλευση και δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την άδεια διερεύνησης ενός κοιτάσματος με την άδεια εξόριξης μελλοντικών ενδεχομένων κοιτάσματων. Επίσης, ε, ε, επαναλαμβάνω, δεν έχει διαπιστωθεί καμία παραβίαση ούτε κανονισμού ούτε οδηγίας και συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας περιμένουμε. Η εταιρεία έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Είναι καθοδόν οι εκθέσεις, δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Άλλος ισχυρισμό για τους οικοτόπους διαφόρων ειδών. Ε, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει καμία παράβαση. Θα γίνει αυτή η μελέτη και η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα δούμε κατά πόσον υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. τα ίδια ισχύουν και με την οδηγία του 2042. Δεν έχει εδώ άμεση εφαρμογή αυτή με τον τρόπο που αναφέρθηκε. Μεταξύ άλλων διότι σε αυτή την περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό. Οπότε Ούτε η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα φύγεται. Υπάρχει μια θαλάσσια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιφορτιστεί με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος για να δούμε ε, πώς θα φτάσουμε στον τελικό μας στόχο και να είναι καθαρές και παραγωγικές οι θάλασσές μας. Όλα αυτά λοιπόν Όλες αυτές οι οδηγίες και τα λοιπά θα συμπεριληφθούν στη μελέτη αντικτύπου που δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί και θα τα λάβει όλα υπόψη. Για μένα είναι απολύτως θεμητές και αξιόπιστες όλες αυτές οι τοποθετήσεις, τεχνικοί, εμπειρογνώμονες που είδαμε ε, και στο βίντεο. Και η Μαρίσα Τεχεδόρ, που ήταν ε, μαζί μου στέλεχο στην πολιτική ζωή και ε, στην τοπική κυβέρνηση των Καναρίων. Τώρα έχει αφοσιωθεί σε άλλες δραστηριότητες. Αλλά όλα αυτά που ακούσαμε είναι καλά επιχειρήματα που ευσταθούν, αλλά πρέπει να τα αναλύσουμε. Όλες ανεξαιρέτως όμως οι παρεμβάσεις και όλα τα επιχειρήματα είναι για το τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχήματος. Τα πουλιά θα πάθουν από το πετρέλαιο γιατί δεν θα μπορούν να πετάξουν, θα έχουν μολυφθεί τα θερά τους. Εντάξει, όλα αυτά που λέτε συνδέονται με ένα πιθανό ατύχημα. Γεγονό είναι ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα να υπάρξει ένα ατύχημα, αλλά είναι μικρές οι πιθανότητες. Και γι' αυτό θα πρέπει να τις ελεγχιστοποιήσουμε και να τις βάλουμε στο πλαίσιο αυτό με διορθωτικά μέτρα και μέτρα πρόληψης. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Έγινε λόγος για πλήρη και απόλυτη πολιτική απόρριψη. Είναι γεγονός ότι τώρα έχει ανέβει πολύ το θέμα. Είδα και πολλά βίντεο. Θα σας πω τα εξής δύο μόνο. Και σε σχέση με τα Κανάρια. 1 1η Φεβρουαρίου 2011, ομιλία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ε, γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος των Καναρίων. Το Κανάριο Σοσιαλιστικό Κόμμα, λέει, ε, με κλειστά τα μάτια θα έκανε τη διερεύνηση. διερεύνηση. Οι μελέτες για την εξόριξη υδρογοναθράκων είναι μόνο θετικές για τα νησιά. Σε άλλη εφημερίδα δεν κατανοώ γιατί αντιτίθεστε με τη διερεύνηση. Έχει ε, πλεονεκτήματα. Ποιο τα λέει αυτά, Γενικό Γραμματέα των Καναρίων Σοσιαλιστών, σήμερα αντιπρόεδρο τη τοπική κυβέρνηση. Άλλε δηλώσει, της ε, συμμαχία των Καναρίων Κοαλισιόν Κανάρια έλεγε ότι βασικός, η ε, βασική πηγή ρήπασης δεν είναι οι πετρολοκυλίδες στα Κανάρια, είναι ο τουρισμός, καταλαβαίνετε τι εννοεί ε, ο έτερος ε, εταίρος της κυβέρνησης. Ήταν και στο εκλογικό τους πρόγραμμα της Συμμαχίας και Συνασπισμού των Καναρίων που σήμερα είναι ο τοπικός Πρωθυπουργό. Ήταν θέμα τους αυτό να διερευνηθούν τα κοιτάσματα ανθράκων που είναι μεγάλου ενδιαφέροντος για το μέλλον των νησιών μας. Αυτό λέγεται κολοτούμπα. Άλλα λέγαμε χτε, άλλα λέμε σήμερα. Ωραία αυτά είναι τα θέματα πολιτικά, τεχνικά, να δημαγωγούμε και να λαϊκίζουμε λυπάμαι και μου κάνει εντύπωση ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στη διερεύνηση που κάνει το βασίλειο του Μαρόκου. Ψυχή ηχθείως, αυτή δεν είναι επικίνδυνη. Και αυτή η δημόσια διαβούλευση, να μην μου πείτε ότι έγινε νυχτιάτικα ή καλοκαιριάτικα. Όταν ανοίγουν προθεσμίες, υπάρχουν, είναι 30 ημερών και μάλιστα διευρύνθηκε η προθεσμία και έγινε 45 μέρες για να μπορέσουν οι πάντες να αντιδράσουν. Και απόδειξη είναι ότι είχαμε 11.000 και κάτι ε, ανθρώπους που διαφώνησαν, εκ των οποίων 5.169 το έκανα γραπτός. Εμένα δεν με πειράζει, ωραία. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το μέλλον, αυτό που είναι σαφές είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα ε, ότι δεν θα συμβούν όλα αυτά και να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ κύριε Μάτο. Κοιτάξτε, βοηθήστε με τώρα τον Πρόεδρο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εγώ δεν έχω και κανένα πρόβλημα να μείνω εδώ και την ώρα του φαγητού. Αλλά έχουμε πρόβλημα. Κύριε Ρωμέβα, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο το αεροπλάνο μου έφταιγε, άκουσα όμως το τέλος και φυσικά γνωρίζω το θέμα γιατί το έχω παρακολουθήσει και επί τόπου ε, και είχα ευκαιρίες επανειλημμένα. Έχω πολλά επιχειρήματα να πω. Πρώτον, χαίρομαι βεβαίως για την υποστήριξη των σοσιαλιστών στο θέμα αυτό και μεταξύ άλλων διότι καταλαβαίνω ότι θα είναι το μοντέλο που θα έχουμε και σε άλλα θέματα και σε άλλες ακτές, έτσι, στην Ισπανία, αλλού στην Ευρώπη, αλλού στον κόσμο. Και χαίρομαι για αυτή τη στάση των σοσιαλιστών. Επίσης, άκουσα και τον κύριο Μάτο και κατανοώ τη θέση του από τη σκοπιά του. Για μένα έχουν σημασία πέντε στοιχεία. Πρώτον, η συμμετοχή δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση όταν μιλούμε για κοινοτική νομοθεσία και ιδιαίτερα για την οδηγία για την ενημέρωση και διαβούλευση του πληθυσμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμμετοχή όταν πρόκειται απλούστατα για ενημέρωση και μάλιστα μεροληπτική του κόσμου χωρίς να υπάρχει διαβούλευση. Δεν ακούνε ε, αυτά που λένε 5.000 πολίτες, το, το είπε ο κ. Μάτο, δεν το λέω εγώ, που έχουν αμφιβολίες. Συμμετοχή δεν σημαίνει απλώς να σε ενημερώσω, θα σου εξηγήσω τι θα κάνω. Ε, συμμετοχή σημαίνει από κοινού να οικοδομήσουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που ε, βραχή, μέσω και μακροπρόθεσμα θα έχει επιρροή ε, στην κοινωνία, στην οικονομία, στο περιβάλλον. Εγώ αλλιώς την αντιλαμβάνομαι τη συμμετοχή, όχι απλώς ενημερώνω για το τι θα κάνω. Και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου επανειλημμένα προσκρούσαμε στην συνήθη πολιτική του συγχρόνου καπιταλισμού. Ε, ιδιωτικοποιώ το κέρδος και κοινωνικοποιώ ε, τη χασούρα, τις απώλειες. Τελικά ποιος πλήρωσε την ύφη, πάντα οι πιο αδύναμοι και εκείνοι που είχαν το λιγότερο λόγο στο κάθε θέμα. Αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Έγινε λόγος για τον κόλπο του Μεξικού. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε. Ξέρουμε τα θέματα. Δεύτερο στοιχείο σημαντικό από τα πέντε που σας είπα είναι η ενεργειακή συζήτηση. Η πιο πολεμοχαρής κυβέρνηση κατά των ανανεώσιμων πηγών ε, ενέργειας, κατά ε, ε, της επένδυσης κεφαλαίου μέσων κτλ συνεχίζει να ποντάρει στην εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και υδρονογοναθράκων. Υπάρχει ένα λάθος στην όλη σύλληψη για το τι ενεργειακό μοντέλο χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, στην Ισπανία και ακόμα περισσότερο στα Κανάρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια θέση από πλευρά του Επιτρόπου Οέτιγκερ και άλλη θέση κάπως διαφορετική από πλευράς των εκπροσώπων του περιβάλλοντος. Αλλά για μένα θα πρέπει να προέχει κυρίως στα, στο μυαλό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο μετασχηματισμός και στα ενεργειακά όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα διάφορα κράτη-μέλη. Το είπε και ο συνάδελφος Λόπες Αγγιλάρ, το θέμα του ανταγωνισμού. Δεν είναι η μόνη περίπτωση όπου ο Υπουργός Βιομηχανίας ευνοεί σαφέστατα ένα πολύ συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μια εταιρεία με πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Και αυτό να το πούμε και κάπως να μας ε, μπουν ψήλοι στα αυτιά. Τέταρτο στοιχείο. Υπερβαλλοντικές επιπτώσεις. Εκτός από πιθανές είναι και ανεπανόρθωτες οι συνέπειες. Αυτό δεν θα πρέπει καθόλου να το υποτιμούμε και ποτέ. Μεταξύ άλλων, γιατί αν θα έπρεπε κάτι να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αρχή της προφύλαξης κάποια στιγμή. Φτάνει πια να γκρινιάζουμε κατόπιν εορτής ότι α, δεν είχαμε χρόνο, δεν είχαμε μέσα να το προβλέψουμε. Πολύ συγκεκριμένο και άμεσο αποτέλεσμα που αφορά τι ακτέ τη Μεσογείου. Ε, το πρόγραμμα ε, του φυσικού αερίου γεωλογικά ε, είναι πολύ ε, ασταθής η περιοχή και ε, είναι πρόβλημα. Και ένα τελευταίο που για μένα δεν είναι ίσονο σημασία, αλλά το σημαντικότερο. Ζούμε σε περίοδους κρίσης και αναζητούμε ad hoc λύσεις από την κρίση. Ο καθένας για να ξεπεράσουμε και κοινωνικά και οικονομικά αυτή την κατάσταση ε, δεινής οικονομίας. Στα Κανάρια νησιά από ό,τι φαίνεται είναι σαφές ότι ο πλούτος που έχουν αυτά τα νησιά είναι να αναπτύξουν τον τουρισμό με νέο τρόπο, με διαφορετικό. Καμία σχέση, καμία όμως σχέση με τη διερεύνηση κοιτασμάτων πετρελαίου που είναι κατά της ποιότητας όχι μόνο του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και ε, θέτει σε κίνδυνο το ε, ίδιο το συμφέρον ε, πολλών και επενδυτών που ποντάρουν και επενδύουν στον τουρισμό που είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία στο νησί. Και τα γνωρίζει πολύ καλύτερο ο συνάδελφο Μάτο. Αυτά και τελείωσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκασές. Και πρέπει να μιλήσω κι εγώ λιγάκι, σας παρακαλώ, να τηρούμε τους χρόνους μας. Ναι, ναι, ναι, σε είδα. Μετά τον Γκαρσές. Εγώ δεν θα επαναλάβω όλα αυτά τα επιχειρήματα που ακούσαμε ήδη. Βεβαίω να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να αναφερθώ σε κάποια θέματα που ακούσαμε. Πρώτον, σε σχέση με την άδεια που έδωσε το 2001 η Ισπανική κυβέρνηση για τη διερεύνηση πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου. Ξέχασε να πει ο ότι το 2004 ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο αυτές οι άδειες. Καλό είναι να το λέμε και αυτό, όχι ότι παρατείνεται η άδεια. Ε, το λησμονήσατε να το αναφέρετε αυτό το στοιχείο και επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό το νομικό στοιχείο. Ακούστηκε και το Μαρόκο. Προς στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πει τίποτα στην κυβέρνηση του Μαρόκου. Καταρχήν, δεν ξέρω, μπορεί από άλλες ε, διαστάσεις και διάβλους να έχει την ευκαιρία κάπως να επηρεάσει αλλά στα χωρικά τους ύδατα που κάνουν εκείνοι ε, αυτές τις διερευνητικές γεωτρήσεις μπορεί να είναι μια συζήτηση πολύ πιο βαθιά για το σε ποιον ανήκουν και οι φυσικοί πόροι. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διάσταση. Απλώς να περιοριστώ στο εξή. Προς στιγμή δεν είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπαγορεύει στην κυβέρνηση του Μαρόχου τι θα κάνει και πού θα διερευνά για πετρέλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όμως μια υποχρέωση να πει κάτι σε μια ευρωπαϊκή επικράτεια όπως είναι οι Κανάριες νήσι. Αυτό μας απασχολεί και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα εδώ. Υπό την κοινοβουλευτική μας ιδιότητα, εμείς ευρωβουλευτές είμαστε και το οφείλουμε σε εκείνους που μας έχουν κλέξει και στείλει εδώ που είναι οι Ισπανοί πολίτες. Με προκειμένο Κανάρι και μαζικά μέσω των θεσμών των τοπικών και των περιφερειακών ήδη έχουν αποβανθεί. Μαζικά, επαναλαμβάνω, κατά αυτών των διερευνητικών ε, γεωτρήσεων ή των αδειών που πρόκειται να δοθούν. Και δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό, να το παραγνωρίζουμε. Έχει κάθε δικαίωμα ο λαός των Καναρίων να εκφράζεται κατά, όπως και έκανε αυτό. Και εμείς ως Ευρωβουλευτές και οι Ισπανοί θα πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ αυτά που λέγει ο λαός των Καναρίων. Μπορεί να τα διαπόψεις από περίσταση σε περίσταση, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σοφό να ε, επανορθώνει κανείς και καλό είναι όταν έχει μια εσφαλμένη άποψη κάποιος και καταλάβει ότι είναι λάθος να επανορθώνει. Και αυτά που μας είπατε δεν ξέρω αν είναι προϊόν παραπληροφόρησης ή ελλειπούς πληροφόρησης. Αξίζει λοιπόν τον κόπο, και εδώ απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν να μην περιορίζεται στην πεπατημένη ή στα τετελεσμένα γεγονότα ειδικά όταν είναι αναφορές τόσο στοιχειοθετημένες και τεκμηριωμένες, να είναι λίγο πιο πολεμοχαρής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή Αναφορών, τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω, θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση που λέγει ότι θα πρέπει να παραμείνει βεβαίω ανοιχτή η αναφορά ή αναφορές, αλλά αξίζει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει και να ζητήσει τις πληροφορίες αυτές που ακόμα δεν γνωρίζει. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να διαβιβάσει και στις αρχές, στην Ισπανική κυβέρνηση δηλαδή, αυτή την απέτηση. Να μην ληφθούν μέτρα και να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αποφευθεί να τεθεί σε κίνδυνο η περιοχή των Καναρίων νησιών και των κατοίκων και κινδυνεύουν δηλαδή να χάσουν όχι μόνο την πηγή της οικονομικής ζωής όπως είναι ο τουρισμός αλλά εκτός των αυτών και επιπλέον και πολύ πιο σημαντικό ίσως από αυτό είναι να μην χάσουν η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλληλεία και οι ίδιοι άνθρωποι το πόσιμο νερό τους εκεί. Θα πρέπει να υπάρξει μια ειφορία και στο χρόνο και στις δραστηριότητε. Παρακαλώ λοιπόν στα συμπεράσματά σας να επιμείνετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεπεράσετε ε, το γνωστό δρόμο που ακολουθήσατε μέχρι τώρα, να επιμείνετε στις πληροφορίες και να αναλάβετε πρωτοβουλίες για να αποφευθούν οι μεγάλοι κίνδυνοι που έχουν καταγγελθεί εδώ και με τους οποίους συμφωνώ απολύτως. Επαναλαμβάνω να παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιράτσα Παΐτια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους αναφέροντες που μας δίνουν την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό που έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία και τεράστιο σάλο. Έχουμε ακόμα 15-16 αναφορές που δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε εδώ και μερικές άλλες που έχουν χαθεί στους δεδάλους της γραφειοκρατίας τη Ζούλη Βενικότ και ο Χωσέ Φινμά και καμιά δεκαριά άλλη ακόμα. Είναι πάρα πολλέ αναφορέ. Εγώ θα επιμείνω στο εξή εδώ. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Δεν με ενδιαφέρει η συζήτηση για τις οδηγίες, αν τηρούνται ή όχι. Υπάρχει πιο βαθύ θέμα, τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, το δικαίωμα των πολιτών του Λανσαρότε και της Φουαρτεβερτούρα να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Το θέμα είναι εμείς τι ε, υπερασπιζόμαστε ιδιωτικά συμφέροντα μιας επιχείρησης για το κέρδος τους ή ε, τα δικαιώματα και το ενδιαφέρον και το συμφέρον των πολιτών. Βεβαίως των πολιτών, αυτό μας ενδιαφέρει μας και όχι τα συμφέροντα των εταιριών. Αυτή η επιτροπή μας εδώ αναφορών θα πρέπει να προασπίσει το δικαίωμα πρόσβαση στο πόσιμο νερό των πολιτών του Λανσαρότε και της Φουερτεβεντούρα. Δεν μπορούμε, λοιπόν να είμαστε υπέρ της διερεύνησης για πετρέλαιο στα ε, χωρικά ύδατα των νησιών αυτών. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη συζήτηση αν παραβιάζονται ή όχι οδηγίας. Θα πρέπει να μπούμε στο βάθος αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι και όχι ε, μεροληπτικά κάποια συμφέροντα. Συμφωνώ με τον συνάδελφο το σοσιαλιστή και το πράσινο εδώ σύντροφο μου να παραμείνει ανοιχτό το θέμα και μας ενδιαφέρει το θέμα των πολιτών και η πρόσβασή του στο δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μέγερ που είμαι εγώ, αλλά ε,